Ladies Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Πρώτη μας συνεδρίαση της χρονιάς. Εύχομαι λοιπόν ό,τι καλύτερο για το 2019 και προσωπικά και σε όλους μας με καλή επιτυχία στις ευρωεκλογές 23 με 26 Μαΐου. Πρώτο σημείο ημερήσια διάταξη έγκριση και έχω κάποιες παρατηρήσεις. Στο σημείο 4 καταρχάς, κατάσταση των σχέσεων Ευρωπαϊκή Ένωση Ρωσία πάει στην αυριανή συνεδρίαση το απόγευμα, 4.30 συγκεκριμένα μετά των Υπουργό Εξωτερικών της Ρουμανίας, θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Κάποια προβλήματα είχε η συγγήτρια, κυρία Κανιέτε, στο πρόγραμμά τη και χρειάστηκε να το αλλάξουμε. Ο κύριο Κόμπια επίση, ειδικό απεσταρμένο για το Αφγανιστάν, έχει κυρώσει την συμμετοχή του αντικαθίσταται από την κυρία Πάολα Παμπαλώνη, αναπληρώτρια ε, Διευθύντρια για την Ασία και τον Ειρηνικό από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και βέβαια το θέμα θα είναι σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν. Εάν δεν έχετε σχόλια ή αντιρρήσεις, εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Σημείο 2. Δεν έχω ανακοινώσεις. σημείο 3. Αν δεν έχετε σχόλια να καταθέσετε μέχρι το τέλος της τρέχουσας συνεδρίας, τα πρακτικά της 29ης, 30 Αυγούστου, 12ης Νοεμβρίου και 26ης Νοεμβρίου εγκρίνονται. Σημείο 4. Επανεξέταση της ε, έκθεσης για την ε, σύσταση της Αντιπροέδρου σχέση με τη στρατηγική επικοινωνία, όπως δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο, και τις σχετικές δραστηριότητες που προγραμματίζονται στο τομέα αυτό. Πλησιάζουν οι ευρωεκλογέ. Καθιστάμεθα όλο και περισσότερο στόχοι ψευδών ειδήσεων, προπαγάνδας, που στόχο έχει να αποδυναμώσει την Ένωση και έτσι Πρέπει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συνεργαστούμε, να ενισχύσουμε την ενθεκτικότητα τη δική μας αλλά και των πολιτών και των γειτονών μας στην αντιμετώπιση αυτής της ε, ψευδούς πληροφορίας. Συστάσεις λοιπόν. Και τώρα δίνω το λόγο στον Τσάρλ Στάνακ, ο οποίος θα μας παρουσιάσει την έκθεση στο όνομα της κυρίας Φωτίγκα. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η κυρία Φωτίγκα ζητεί συγγνώμη. Για λόγους υγείας δεν μπόρεσε να έρθει σήμερα. Την αντικαθιστώ λοιπόν την αντικατάσταση μάλιστα και κατά τη διαπραγμάτευση των συμβαστικών τροπολογιών την προηγούμενη εβδομάδα. Και έτσι την εκπροσωπώ. Είχαμε σκιώδεις εισηγητές, εξαιρετικά έμπειρους. Μαζί τους λοιπόν προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κληθεί μαζί με τα άλλα θεσμικά όργανα να αναπτύξει περισσότερο τι δραστηριότητε του στην ε, αντιμετώπιση των εχθρικών αυτών επιχειρήσεων παραπληροφόρηση. Καλούμε εδώ και τα κράτη-μέλη να αξιολογήσουν το καθένα στην επικράτειά του την κατάσταση. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία ζητεί να δοθεί στην προτεραιότητα στο θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτείνει μια σειρά από για την μεταβολή το εις προσέγγιση των θεσμικών οργάνων, το συντονισμό των δράσεων, την αντιμετώπιση των ζητημάτων τεχνητής νοημοσύνης και νέων τεχνολογιών και μέτρων αντίστοιχων για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής. Θεωρούμε ότι μια εις ανάλυση και έρευνα για τις επιπτώσεις και τον αντίκτυπο εχθρική προπαγάνδας είναι απαραίτητη προκειμένου να αναπτυχθούν μέτρα που θα ε, αντιμετωπίσουν επιτυχώς αυτούς τους κινδύνου. Θεωρούμε πάντως και το δηλώνουμε εξ αρχή ότι η ελευθερία του λόγου, της έκφραση και του τύπου ε, είναι στο επίκεντρο κάθε δημοκρατικής κοινωνίας. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία σε όλη την έκθεση σε όλη τη διάρκεια τη επεξεργασία τη και της διαπραγματεύσει για τις συμβαστικέ τροπολογίες. Ελπίζω δε ότι το κείμενο όπως έχει τροποποιηθεί κατά την αυριανή ψηφοφορία θα εγκριθεί. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Τσόλ Στάνοκ. Και οι συνάδελφοι τώρα, ποιο θέλει να λάβει το λόγο, οι οπωσδήποτε πρώτα. Παρακαλώ, η κυρία Μανέσκου Ελκ. Σα Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ θερμά την κυρία Φωτίκα για το έργο της και όλους του κοιόδη ηγητές για την ε, συνεργασία που είχαμε. Συμφωνήσαμε για 27 συμβαστικέ τροπολογίες και νομίζω το κείμενο που προέκυψε είναι καλό, γιατί αναγνωρίζει την ύπαρξη τέτοια προπαγάνδας και την ανάγκη προορατικών μέτρων προκειμένου να καταπολεμηθεί, να αντιταχθούμε σε αυτή την εχθρική προπαγάνδα και φυσικά εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Και ενώπιση των ευρωεκλογών θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον υβριδικό πόλεμο και την παραπληροφόρηση. Γιατί ήδη έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από τότε που το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε αποτελεσματική αντίδραση στην εξτρατεία παραπληροφόρηση που οργάνωσε η Ρωσία. Και επιτέλους μπορούμε να πούμε ότι είναι όρατες, προβεβλημένες και αποτελεσματικές οι δράσεις μας, γιατί έχουμε τη online πλατφόρμες και ένα δεντολογικό κώδικα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της παραπληροφόρησης. Και πέρυσι το Δεκέμβριο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε και ένα σχέδιο δράσης με κατάλληλα και ακριβή μέτρα για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να εφαρμόσουμε αποτελεσματικά αυτό το σχέδιο δράσης γιατί σίγουρα ε, λόγω των επικείμενων ευρωκλογών ε, είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε επιτυχία στην ε, εκστρατεία μας για να επαναφέρουμε την ε, βεβαιότητα, την εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και ευελπιστώ ότι θα έχουν ο πέρας οι συζητήσεις της έκθεσης Φωτίγκα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φρόιντ από τους Σοσιαλιστές. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα ξεκινώντας να ευχαριστήσω βεβαίως και εσάς κύριε Πρόεδρε για την επισκόπηση όλου του ζητήματος που μας παρουσιάσατε και βεβαίως δεν θα τα αναπτύξω πάλι όλα, αλλά ιδιαίτερος και τον Τσάρλ ε, Στάνοκ ο οποίος απεδείχθη πολύ επιτυχής διαπραγματευτής κατά τις ε, συνομιλίες των σκιωδών. Και ιδιαίτερος βέβαια ευχαριστώ, ευχόμενος και από τη θέση αυτή ε, ταχεία ανάρρωση, την αγαπητή Φωτίνκα. Το σχέδιο έκθεσης είναι νομίζω και μπορούμε να το πούμε έτσι μια ε, αυτονόητη συνέχεια της έκθεσης που είχαμε το 2016 για την καταπολέμηση της ανετικής της ψεύδους προπαγάνδας, της έκθεσης δηλαδή για τη στρατηγική επικοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την, ε, για την αντιμετώπιση προπαγάνδας που απευθύνεται εις βάρος της αποτρίτους. Δηλαδή ψευδείς ειδήσει, ε, παραπληροφόρηση, προπαγάνδα κτλ. αντιμετωπίστηκαν με μια πληθώρα μέσων. Τώρα λοιπόν έχουμε προτείνει μια σειρά από που αντιστοιχούν σε προκλήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να δουν την ανάπτυξη στοχευμένων εκστρατιών αντιμετώπισης της προπαγάνδας με τα, κοινωνικά μέσα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δηλαδή, αλλά και με την κοινωνία των πολιτών που μπορεί να ε, λάβει μέρος σε αυτή τη δύσκολη επιχείρηση. 25 ή 26 ήταν οι συμβαστικές τροπολογίες και πιστεύω ότι μετά το, την τελική ψηφοφορία θα έχουμε ένα καλό έγγραφο, ένα έγγραφο το οποίο θα δίνει αποφασιστική απάντηση στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ε, ε, εκστρατεία παραπληροφόρηση και ψευδών ειδήσεων. Ξέρουμε ότι πολλά από αυτά προέρχονται από τη Ρωσία, το έχουμε διαπιστώσει και το έχουν επισημάνει και πολλοί, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχουν και θέλουμε ιδιαίτερα να δώσουμε έμφαση στο γεγονό ότι υπάρχουν και άλλα κράτη, η Κίνα, η Βόρεια Κορέα, το Ιράν, που αναπτύσσουν τέτοιου είδου ε, επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και επίσης με ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογία ε, υπηρεσίες σε παραδείγματι messenger ε, μηνυμάτων αλλά και ο τομέα τη τεχνητής νοημοσύνης που βλέπουμε ότι μπορεί να παρασυρθεί σε αυτή την αρνητική εκστρατεία. Και επιπλέον θα ήθελα, ευχαριστώντας και τον πρόεδρο που το ανέφερα, να τονίσω πως ο χρόνος πιέζει, έχουμε, έπονται οι ευρωεκλογές, πολύ γρήγορα θα έρθουν και θα δούμε εξελίξεις οι οποίες πολύ φοβάμαι ότι θα είναι στην ευρύτερη έννοια της λέξης αντιπαραγωγικές για το δημοκρατικό γίγνεσθε. Ο πρόεδρος ευχαριστώ πολύ, ο Ίγκεν Φρόεντ, από τους φιλελεύθερους Πέτρας. Thank Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να στείλω τις ευχαριστίες μου μέσω του Charles Τάνοξ στην Άννα Φωτίγκα για την αγαστή συνεργασία που είχαμε, το εξαιρετικό της έργο και για το γεγονός ότι επιμένει στην προτεραιότητα αυτή. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους συναδέλφους, τους παρόντες τουλάχιστον, ότι το 2016 είχαμε την τύχη να συντάξουμε την πρώτη έκθεση για την ε, προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Τότε είχε σοκάρει πολλούς ε, και δεν συμφωνούσαν όλοι με την ύπαρξη, την παρουσία της εχθρικής προπαγάνδας κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εταίρων της. Αλλά η πραγματικότητα αυτή είναι δεδομένη πια τη ύπαρξη τέτοια εχθρική προπαγάνδας Και ελπίζω να τύχει ευρεία υποστήριξη αυτή η έκθεση στην αυριανή μας ψηφοφορία. Θα ήθελα να σταθώ σε τρία σημεία που κατά τη γνώμη μου συνιστούν σαφή πρόοδο σε σχέση με την πρώτη σχετική έκθεση του 2016. Καταρχήν, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο, σαφέστατο μήνυμα και στοχευμένες δράσεις και κυρώσεις ε, των δραστών αυτής της συνορχιστρωμένης εχθρικής ε, προπαγάνδας και της παραπληροφόρησης. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα της επιβολής κυρώσεων, στοχευμένων κυρώσεων. Κάτι που θα είναι ένα πολύ κατάλληλο αποτρεπτικό μέτρο. Όχι να μιλά κανείς για προπαγάνδα και παραπληροφόρηση, αλλά να ενεργοποιηθούν και όλα μερικοί για να αποτρέψουν τους δράστες από την διάπραξη τέτοιων ενεργειών παραπληροφόρηση και εχθρικής προπαγάνδας. Δεύτερον, χαιρετίζουμε την σύσταση τριών ομάδων εργασίας για την Ανατολική Ευρώπη, τα Δυτικά Βαλκάνια και το Νότο. Τρεις ομάδες εργασίας, τρεις ομάδες κρούσης που καλύπτουν ε, ε, μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Ανατολή, Βαλκάνια και Δύση και Νότο. Και σίγουρα θα πρέπει να στηρίξουμε αυτές τις τρεις ειδικές ομάδες εργασίας και να ε, συνεπικορίσουμε στο τεράστιο έργο που έχουν να επιτελέσουν. Επίσης, είναι προτεραιότητα του επόμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της είπα της εκπροσώπου να εξασφαλίσουν επαρκείς πόρους και τους κατάλληλους μηχανισμούς ώστε πραγματικά να έχουμε μια δέσμη μέτρων, ένα πλούσιο πλωστάσιο για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Πιστεύω αγαπητοί συνάδελφοι ότι η έκθεσή μας, η έκθεση Φωτίγκα θα στηρίξει και θα προωθήσει τις, ε, την έκκλησή μας για σωστές στρατηγικές και τονίζουμε την ανάγκη να καταπολεμήσουμε την παραπληροφόρηση και την εχθρική προπαγάνδα, που δεν είναι καθόλου θεωρία. Είναι πραγματικά μια πρακτική που θα τη διαπιστώσουμε και στη διάρκεια των ευρωεκλογών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον Πέτρα Σταστρεβίτσιος και από τους πράσινους τώρα η Ρεμπέκα Χάρμς. Ναι, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Τσάρλς Στανάκ ο οποίος ε, με λίγο χρόνο στη θέση του και με πάρα πολύ ικανοποιητικό τρόπο οργάνωσε και καθοδήγησε τις εργασίες των σκιωδών ε, και η κυρία Ποτίγκα βεβαία, αλλά και ο κύριος Αουστρεβίτσος ε, και θα συμφωνήσω μαζί του ότι ήταν πολύ χρήσιμο για την έκθεση αυτή το γεγονός ότι όλοι μας έχουμε συλλέξει πολύ περισσότερη εμπειρία στο διάστημα που έχει παρέλθει με, σε σχέση με μη φιλικές ή ακόμα λιγότερο φιλικές δράσεις προπαγάνδας σε σχέση με τη Ρωσία. Και βεβαίως και το θέμα της ε, εμπλοκής της στην εκστρατεία του Brexit και για τη δουλειά που έχει κάνει στην εκστρατεία του Τραμπ στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε υπόψη και στη γερμανική μάλιστα εκλογική διαδικασία μπορέσαμε να δούμε ίχνη αυτή τη εμπλοκή τη Ρωσίας και νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε και τη συνέχεια στην επικυρότητα με την ε, έμφαση που δίνουν μέσα ε, ενημέρωσης ρωσικών συμφερόντων ή επίδρασης, επιρροής, ε, στην έμφαση λοιπόν που δίνουν στο κίνημα των κίτρινων γυλαίκων τη σύγχρονη εποχή αυτές τις μέρες. Και νομίζω ότι μπορούμε να δείξουμε ως Κοινοβούλιο και περισσότερη φιλοδοξία και να κάνουμε ε, να δώσουμε καθαρά επιχειρήματα απέναντι σε αυτήν την ε, προπαγάνδα. Προσπαθώντας βέβαια να μην ξεπεράσουμε αυτή τη λεπτή γραμμή που μας ξεχωρίζει από την αντιπροπαγάνδα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή η γραμμή να είναι σαφής. Γιατί με μια αντιπροπαγάνδα δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την μη φιλική ή εχθρική ε, προπαγάνδα. Μπορούμε όμως με την εξήγηση, με την ενημέρωση, με την αποκατάσταση της αλήθειας, με ποιοτική δημοσιογραφία, με ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να κάνουμε πολύ περισσότερα από όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έρχεται στην κατάλληλη στιγμή λοιπόν αυτή η έκθεση και μάλιστα και η επίτροπο Γιώροβα με την πρωτοβουλία τη να οργανώσει μεταξύ κρατών μελών και ε, Βρύξελων συζήτηση για το θέμα αυτό ενώπιση των ευρωεκλογών νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει και πολύ σημαντική υποστήριξη στο έργο Μα. Ευχαριστώ λοιπόν για τη συνεργασία και ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Στάνοκ που ε, τόσο, μέσα σε τόσο σύντομο διάστημα ανέλαβε ε, την καθοδήγηση των εργασιών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόσο, τελευταίος. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ήδη είχαμε ψηφίσει κατά της έκθεσης όταν εγκρίθηκε από την Ολομέλεια, όπου είχαμε και μεγάλη αποχή, για παράδειγμα, από τους σοσιαλιστές. Και θα θέλαμε να είχαν ψηφίσει όπως εμείς, γιατί βλέπουν υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα. Καταρχήν, θέλουμε περισσότερες προφορίες για το τι ακριβώς είναι η παραπληροφόρηση και τι είναι η προπαγάνδα. Αυτό που μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η πιθανότητα αυτός ο κοινοτικός μηχανισμός να μας οδηγήσει σε λογοκρισία ή σε αυτολογοκρισία τους δημοσιογράφου, κάτι το οποίο θα επηρεάσει αρνητικά ε, το όλο κλίμα της συζήτησης που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε τελείως κατά πρωτοβουλειών οι οποίες θέλουν να επιβάλλουν κυρώσεις σε δημοσιογράφους και τι περίεργο αυτό προέρχεται από τους φιλελεύθερους. Πρέπει να σας πω πως δεν έχουμε απόλυτα τεκμήρια που να αποδεικνύουν πως είχαμε παρέμβαση της Ρωσίας ε, που να επηρεάζουν τις εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη ΣΥΠΑ. Ξέρουμε πως ε, η κυρία Χάρ προσπαθεί να με ε, διακόψει. Είναι φοβάται τη Ρωσία, αλλά δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο. Και αν ε, το εκλογικό σώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να τιμωρήσει κάποιες ε, κυβερνήσεις, αυτό έχει να κάνει με το νεοφιλελεύθερο καθεστώς που επιβάλλουμε από τι Βρυξέλλε. Να σας πω τώρα για τις ε, θεωρίες που ακούγονται για τα μίντια. Εμείς που γνωρίζουμε τα τη επικοινωνία. αυτά όλα έχουν ήδη απορριφθεί από το παρελθόν. Δεν είναι τώρα κενές φιάλες οι οι συμπολίτε μας που μπορούν να τι γεμίσουμε με ένα σωρό ψευδεί ειδήσει. Όχι, μόνο όταν υπάρχει γόνιμο έδαφος είναι πετυχημένε αυτές τι προσπάθειες. Και τώρα, μιλάμε για μια συγκεκριμένη χώρα. Ε, λέμε για τη Ρωσία. Αυτή τη στιγμή χειροτερεύουν οι σχέσεις μας χωρί να υπάρχουν απόλυτε αποδείξει για κάτι τέτοιο. Γιατί αναφέρθηκαν πολλέ χώρε και έχουμε και προτάσει από φιλελεύθερου και, και από ε, τους ε, εκπροσώπους του ΕΛΚ είναι Ρωσία, Κίνα, ε, Κορέα, Βόρειος Κορέα, ε, χώρες από τις οποίες φοβούνται οι ΙΠΑ και για τις οποίες προσπαθούν να στρέψουν εναντίον τους το ευρωπαϊκό κοινό. Βεβαίως ε, προήρθαν κάποιες επιθέσεις από εκεί, αλλά για την πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για τις επικοινωνίες οδηγεί σε στρατικοποίηση του χώρου της επικοινωνίας και ανοίγει την πόρτα σε κινδύνους κατά της ελευθερίας ε, σκέψης, επικοινωνίας και πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καταστρατηγεί και τις θεμελιώδει αρχές, τα άρθρα 7 και 8 της Ευρωπαϊκής ε, Συνθήκης. Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο το οποίο μας επιτρέπει ε, να ε, φιλτράρουμε ε, τις πληροφορίες. Ποιο είναι, ποια είναι η νομική βάση που μας επιτρέπει να κινηθούμε κατά δημοσιογράφων. Αυτά θα θέλαμε να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κόουσο. Δύο ακόμα έχουν ζητήσει το λόγο. Αγκόμες και Φλέκενστάιν, άλλος κανείς. Παρακαλώ πολύ, η Άννα Νομίζω πως είναι ξεκάθαρο πως έχουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Και δεν συμφωνώ πως χρειάζεται ορισμός. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ψευδείς ειδήσει, ψευδείς στοιχεία και όπου η πραγματικότητα έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα στοιχεία. Και έχουμε περιπτώσεις όπου η χρήση αυτών των στρεβλωμένων αφηγημάτων της πραγματικότητας οδηγούν σε χειραγώγηση πολιτικών αποτελεσμάτων, το Brexit είναι ένα καλό παράδειγμα, τότε αυτό ναι δείχνει πως όπως είπε και ένας δημοσιογράφος του Guardian και του Observer οδηγούν στο να μπορούν κάποια άτομα τα οποία είναι εγκαταστημένα στη Βρετανική κοινωνία να χρηματοδοτούν και να ε, ε, πετυχαίνουν αποτελέσματα που επιθυμούν. Τι έγινε με την Cambridge Analytica, τι έγινε με τα δεδομένα εκεί. Είναι γελίο που ακόμα αρνιόμαστε να δούμε την πραγματικότητα. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός πω έρευνε σοβαρές που γίνονται από δημοσιογράφου που δεν έχουν δεν, είναι υποκινου... Ε, δεν έχουν υποκινηθεί πολιτικά, ε, μας οδηγούν να το πιστέψουμε. Και γιατί να το αρνηθούμε. Γιατί να αρνηθούμε κάτι το οποίο η κυρία Λεπέν δεν αρνήθηκε. Ότι όντως η δική της εκστρατεία στη Γαλλία χρηματοδοτήθηκε από μια ρωσική τράπεζα η οποία συνδέεται ξεκάθαρα με τον Πούτιν. Αυτό πώς θα το αρνηθούμε. Ούτε ήδη δεν το αρνήθηκαν όταν αποκαλύφθη. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο η Ρωσία, το πήγε κάποιος άλλος, είναι και άλλα καθεστώτα τα οποία έχουν ε, πολιτικές επιδιώξεις οι οποίες δεν ε, συνδυάζονται με ούτε προορισμό ούτε με δημοκρατική έκφραση γνώμεων και βέβαια ναι εδώ θα πρέπει και την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία να τα συμπεριλάβουμε ως κράτη και έχουμε και κάποιους οι οποίοι αγοράζουν πολιτικούς και δεν χρηματοδοτούν απλώς εκστρατείες και κόμματα, αλλά αγοράζουν πολιτικούς έτσι ώστε να τροφοδοτήσουν ένα αφήγημα το οποίο δεν επιτρέπει την ελεύθερη και δημοκρατική έκφραση ε, των ανθρώπων. Δεν μπορούμε να τονιθούμε και γι' αυτό στηρίζω την πρόταση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ο Κνούτ. ναι, ευχαριστώ. Και θέλω να απαντήσω μόνο σε εσάς της ΓΚΟΕ. Δεν ε, ε, θεωρούμε εχθρός της Ρωσίας. Κι αν έχετε κάποια εμβολία, ελάτε αύριο το πρωί και θα αποδειχθεί. Αλλά δεν μπορούμε να αρνούμε αυτά τα γεγονότα. Ακόμα και να λέγαμε άμα δεν είναι μονομερής η θεώρηση, η επιθέση, γιατί και εμείς έχουμε ένα κομμάτι, έχουμε κάποια κομμάτια αυτού του τύπου προπαγάνδας. Δεν θέλω οπωσδήποτε να τα βάλω σε, στο ίδιο επίπεδο, να τα συγκρίνω βέβαια. Μπορούμε να κάνουμε το εξή. Ή να το αρνούμεθα, ή να το δεχόμαστε αρνούμενοι ότι υπάρχει πρόβλημα, ή να καταφύγουμε στην ε, λογοκρισία ή την ε, αντιπροπαγάνδα. Η έκθεση λοιπόν που έχουμε εδώ νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα χωρίς να ζητεί αντιπροπαγάνδα ή άλλα πράγματα που δεν θα θέλαμε. Και γι' αυτό δεν έχω ενδιασμούς να την υποστηρίξω. γιατί νομίζω ότι ούτε στον εαυτό μας, ούτε σε εμά τους ίδιους, ούτε και στη Ρωσία θα κάναμε καλό αν καταλήγαμε στο επιχείρημα Α, από όλες τις πλευρές υπάρχει αυτό και το ίδιο κάνει. Όχι, δεν κάνει το ίδιο. Και πρέπει να αντιδράσουμε. Και νομίζω ότι θα το αναγνωρίσει και η Ρωσία. Ευχαριστώ, Κνούτ. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να σας ενημερώσω για το χρονοδιάγραμμα. Ψηφοφορία 22 Ιανουαρίου στην Επιτροπή μας και στην Ολομέλεια, μάλλον το Φεβρουάριο. Έχουμε λίγο αργήσει. Πάμε στο σημείο 5. Συστάση προ την Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή που Εκπροσωπού τη Ένωση για θέματα εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια σχετικά με τον απολογισμό της συνέχειας κτλ. Και είναι το σημείο 6 της Μερικής σχετικά με τη συνολική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ουσμπεκιστάν. Η συγκητή είναι ο Από το 1999 ισχύει αυτή η συμφωνία. Οι συνομιλίες για τη νέα ξεκίνησαν στις 23 Νοεμβρίου του 2018 Στόχος είναι να διατηρηθεί ο πολιτικός διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφενό και Ουσμπεκιστάν αφετέρου, ενώ συνεχίζονται οι μεταρρυθμίσεις σε κάθε τομέα για την εξασφάλιση σταθερών θεσμών, πολυφωνίας, ε, σταθερού δικαστικού συστήματος υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση και την, ε, το περιβάλλον στη χώρα και Πρέπει να ενθαρρυνθεί το Ουσμπεκιστάν να ενταχθεί στην ε, Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Είχαμε το Σεπτέμβριο του 2018 μια συνεδρίαση με επαφέ που δεν μπόρεσα δυστυχώ εγώ να παρακολουθήσω. Ωστόσο, οι συνάδελφοί μου είπαν ότι σημείωσαν σημαντικέ αλλαγέ, κοινωνικοπολιτικέ εξελίξει με, με σε σχέση με προηγούμενη συνεδρίαση που είχε γίνει το 2015, με τη νέα εξωτερική πολιτική του Σμπεκιστάν που έχει αναπτύξει και την περιφερειακή συνεργασία και έχει συμβάλει και στην ε, διαδικασία ειρηνεύση του Αφγανιστάν. Άλλη θετική εξέλιξη είναι το γεγονό ότι αποφυλακίστηκαν πολιτικοί κρατούμενοι, ότι έχει ε, δικαίωμα ε, πολιτικού ελέγχου του εκτελεστικού το κοινοβούλιο και άλλες αρμοδιότητες λάβει εντωμεταξύ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Παραδείγματι, βέβαια, πρέπει εμεί να επαγρυπνούμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα πάντα και γι' αυτό και αυτή είναι η τελευταία μου παρατήρηση. Ο στόχο τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσφέρει την υποστήριξή τη στο Ουσμπεκιστάν με τι ιστορικέ δημοκρατικέ διαδικασίε αφενό, αφετέρου και τι εξωτερικέ προσπάθειε για το διεθνή, περιφερειακή και παγκόσμια συνεργασία και βέβαια να στοχεύσουμε σε μια πιο ε, φιλόδοξη συμφωνία σε σχέση με την τρέχουσα συμφωνία εταιρικών σχέσεων. Αυτά από μένα οι σκιώδεις ηγητές θα λάβουν το λόγο. Ε, δεν έχει ζητήσει από τους σοσιαλιστές δημοκράτες κανένας, επομένως δίνω το λόγο στον Σαλστανόκ. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια του κ. Τάνοκ. Ε, κανονικά δεν είχα ζητήσει το λόγο και δεν δίνετε το λόγο, είμαι λίγο απροετοίμαστος. Πάντως η έκθεση είναι εξαιρετική θα έλεγα και η ομάδα μου ανέκαθεν ήταν υπέρ ε, των, ε, της σύγκλησης με τις δημοκρατίες της Κεντρικής Ασίας και με το Ουσπεκιστάν ιδιαίτερος ε, για να σφίξουμε τις πολιτικές και εμπορικές μας σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια στο παρελθόν μα προβλημάτιζε η ιδιαίτερη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στη χώρα αυτή και η έλλειψη τη δημοκρατία και η χρήση παιδική εργασία, Αλλά αυτά τα θέματα έχουν ε, ληφθεί υπόψη και επισημαίνονται και στην έκθεση και σίγουρα πρέπει να σφυριλατήσουμε πιο στενού εμπορικούς και πολιτικούς δεσμού, ασκώντα έτσι καλύτερα πίεση στην κυβέρνηση και πιο αποτελεσματικά στην κυβέρνηση της Τασκένδης να βελτιώσει την κατάσταση. Αυτά. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη. Δεν είχα δει από εδώ από την άντρα ότι ο κύριος Μπενιφέ έχει ζητήσει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε πως έχουν αλλάξει οι σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουσμπεκιστάν. Στη διάρκεια μιας μόνο βουλευτικής ε, περίοδου η παλαιά συμφωνία συνεργασίας και το πρωτόκολλο για τα κλωστοιφαντουρκικά, που είχε μάλιστα αρθεί η εφαρμογή του λόγω της εργασίας των ανηλίκων κτλ. Ε, αλλά και η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε σχέση με την ε, διεθνή οργάνωση εργασίας, ε, τη μείωση του, της παιδικής εργασίας. Προτάθηκε λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο χρόνια η αυτής της άρσης εφαρμογής του πρωτοκόλλου μπορούμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με τη μεγαλύτερη χώρα γείτονα του Καζακ... μετά το Καζακστάν και για να συνεχίσω στην, ε, ε, στους παραλληλισμούς αυτούς θα ήθελα να σημειώσω ότι τέτοιου ίδιου σχέσεις ε, βελτιώνουν την αντανάκλαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο παγκόσμιο σκηνικό. Έχουμε να κάνουμε και με την νέα ηγεσία του Ουσβεκιστάν, ιδιαίτερα ο πρόεδρος Μιτζιόιεφ έχει λάβει μια νέα, έχει κάνει νέες επιλογές, διαφορετικές επιλογές σχέσεις και με τα εσωτερικά αλλά και με τις σχέσεις, στις σχέσεις με τις γειτονικέ χώρες, σχέσεις που παραδοσιακά ήταν πολύ τεταμένες. Οι Ουιγούροι στο Τατζικιστάν μέχρι πρόσφατα απειλούσαν ε, να προξενήσουν μια ένα περιφερειακό πόλεμο, μια περιφερειακή σύραξη. Προβλήματα είχαν επίσης με την ε, Αράλη, τη λίμνη Αράλη που αποτελούσε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα, για να μην πω περιβαλλοντική καταστροφή του 21ου αιώνα και αυτό πάλι αντιμετωπίζεται και έχουμε μια πρόοδο ε, περιορισμένη ίσως αλλά σημαντική στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την αποφυλάκηση των πολιτικών κρατουμένων και με την βελτίωση των σχέσεων ε, με τους ε, εκπροσώπους οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μένουν ακόμα θέματα συνδικαλισμού, μένουν ακόμα προβλήματα σε σχέση με τους ΛΟΑΔΜ που θεωρούνται, θεωρείται πως δεν πράττουν ακόμη ποινικό αδίκημα και αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Νομίζω ότι μπορούμε και να σημειώσουμε πως ε, στο θέμα της ε, συλλογής βάμβακα και μέταξας ε, με καταναγκαστική εργασία χρειάζεται ακόμη περισσότερη προόδος πλουραλισμός, χώρος ε, ανάπτυξης δραστηριότητα της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και δικαιοσύνη, όπως και σοφρονιστικό σύστημα είναι προβλήματα ακόμη στη χώρα αυτή και βέβαια και οι προοπτικές της οικονομίας είναι αρκετά ανησυχητικέ. Όλα αυτά τα ε, περιγράφει ικανοποιητικά το καλό κείμενο της γνωμοδότησης και το, ε, ευχαριστώ τον πρόεδρο και εισηγητή μας κύριο Μακάλιστερ. Μια-δυο τροπολογίες θα κάνω για να βελτιώσω κάποια σημεία κυρίως όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Thank you, Σας ευχαριστούμε κύριε Μπενιφέη. Δεν ζητά κάνει το λόγο από τους φιλελεύθερους ή τους πράσινους, οπότε δίνω το λόγο στον κύριο Σόλτς από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά για το σχέδιο έκθεσή σας. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να συζητήσουμε τις σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει μια χώρα που εξακολουθεί να περνά αυτή τη μεταβατική διαδικασία του μετασχηματισμού. Βέβαια, έχουμε διαπιστώσει μια βελτίωση της κατάστασης σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, αλλά ακόμη η κατάσταση δεν είναι πλήρης, ε, τέλεια, γιατί ε, πρέπει να συνεχιστεί η ολοκλήρωση του μετασχηματισμού αυτής της χώρας για να μην μείνει στη μέση. Πάντως συμφωνώ με τους προλαλήσαντες ότι σίγουρα υπάρχουν ε, σημαντικές και αισθητέ επιτυχίες, ε, σημαντικά επιτεύγματα προς μια βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας που έχει τις δικές της βάσεις και γίνονται κάποιες απόπειρες διαφοροποίηση της οικονομίας. Ε, από το παλιό μονοπόλιο του, της βαμβακοβιομηχανίας που ίσχυε στο παρελθόν. Βέβαια, αυτή η διαδικασία μετασχηματισμού του Ουσμπεκιστάν θα πρέπει να συνδεστεί με το πολιτικό σύστημα και την πολιτική ηγεσία που προσπαθεί να κρατήσει την εξουσία στα πλαίσια της ε, ε, ελίτ που διακυβερνά τη χώρα. Και Γι' αυτό, όπω λέτε και στην έκθεση, θα πρέπει να διεκδικήσουμε σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών. Γιατί εκεί υστερεί κάπω η χώρα και είναι σωστό να το επισημαίνουμε. Τέλο, θα ήθελα να επισημάνω ότι στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφή στο Κατοβίτσα για την εφαρμογή τη Συμφωνία των Παρισίων για τι κλιματικέ αλλαγέ, ε, θεωρώ ότι για το Ουσμπεκιστάν ε, ιδιαίτερα η υλοποίηση της προστασίας της ποιότητας του ύδατος και η επαναθεώρηση της χρήσης του ύδατος είναι πολύ σημαντικό για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και είναι και προς το συμφέρον των πολιτών της, αλλά και προς το συμφέρον του περιβάλλοντος. Οπότε πιστεύω ότι θα πρέπει από εκείνο να σκεφτούμε πώς θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη χώρα αυτή, προκειμένου να συνεχιστεί η ανανέωσή της και η ε, περαιτέρω οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική της ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Σόλτς. Δύο ακόμη συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Ο Μίχελ Γκάλερ και η Άννα Γκόμες. Άλλος κανείς? Όχι, οπότε ο κύριος Γκάλερ. Ευχαριστώ για την έκθεση και τη γραμμοδότηση και τους κοιόδης. Βεβαίω την υποστηρίζω. Είχα την ευκαιρία μάλιστα πέρσι να ρίξω μια γρήγορη ματιά στη χώρα Όλα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν εδώ ε, είναι ζητήματα που μας αφορούν σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν. Σημαντικό είναι αυτό τον, της κλωστοϊφαντουργίας και της εργασίας των παιδιών. Ψυχολογικά κιόλα. Είναι πολύ σημαντικό το ότι έχει διευθετηθεί και θεωρούμε πάντως ότι δεν σκοπεύει η κυβέρνηση να συνεχίσει την απασχόληση παιδιών στην κλωστή Θεωρούμε δηλαδή ότι δεν είναι τόσο βασικό πλέον το πρόβλημα αυτό. Δεν ε, επιβάλλεται, ούτε αποκρύπτεται, ούτε γίνεται ανεκτό τουλάχιστον το φαινόμενο της ε, παιδικής εργασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι η άλλη πλευρά ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για συνεργασία μαζί μας ε, και αν ε, συνάψουμε μια νέα συμφωνία τη θεωρούν ευπρόσδεκτη. Εγώ πάντα και με θετικό τρόπο συνέδεα και τις δικές μου θέσεις με αυτές τις ε, προτάσεις του Προέδρου ότι η προσέγγιση θα πρέπει να ακολουθεί όχι μια άνωθεν επιβολή αλλά την εξέλιξη της κοινωνίας και της πολιτικής. Δηλαδή η κοινωνία να θελήσει και να ενστερνιστεί αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις. Θα τα συστήσουμε φυσικά. Είμαι αισιόδοξο πάντως ότι βρισκόμαστε σε σωστό δρόμο. Και άλλωστε νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι ό,τι γίνεται γίνεται για το καλό της χώρας αυτής. Ευχαριστώ τον κύριο Γκάλερη, Άννα Γκόμες. Πήγα πριν από μερικά χρόνια στο Ουσμπεκιστάν, αν δεν κάνω λάθος, το 2008. Και τα προβλήματα με τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν τεράστια. Η ηγεσία ήταν σε απόλυτη άρνηση για τα τεράστια προβλήματα που είχαν και κυρίως το θέμα της παιδικής εργασίας. Φέτος ξαναπήγα με την αντιπροσωπεία της ΑΦΕΤ και είδα πως έχουν γίνει πραγματικές αλλαγές και το γεγονός το ότι πέθανε ένας δεινόσαυρος και απελευθερώθηκε η χώρα, γιατί αυτό έγινε στο Ουσμπεκιστάν. Και είναι μεγάλη διαφορά με τα όσα είδαμε στο Καζαχστάν, την ε, γειτονική χώρα, όπου ο δεινόσαυρος υπάρχει και καταπιέζει. Στο Ουσμπεκιστάν συγκινήθηκα που γνώρισα και πρώην πολιτικούς ε, κρατούμενους οι οποίοι απελευθερώθηκαν και τη διαφορά την οποία οι αισθάνονται. Και όπως είπαν πολλοί συνάδελφοι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι ακόμα πολλά. Είναι όμως διαφορετική η στάση τους. Και εδώ έχουμε το κάθαρο παράδειγμα ε, που έχουμε μια χώρα που δεν χρειάζεται μόνο εξωτερική πίεση, αλλά υπάρχει και μια κατανόηση του ότι είναι προσφέρον της χώρας να ανοίξει, να αποδεχτεί την κριτική και να βρει τρόπους να αντιμετωπίσει τις όποιες επικρίσεις. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποια χώρα στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση με στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στα πλαίσια της σφαιρικής συμφωνίας που διαπραγματευόμαστε ε, είναι ελπιδοφόρο, τότε η χώρα αυτή είναι το Ουσμπικιστάν. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλους ομιλητές στον κατάλογο. Να σας πω λοιπόν πως 23 Ιανουαρίου τροπολογίες, 11 το πρωί. Στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε στις 21 Φεβρουαρίου και θα περάσουμε από τη δεύτερη Ολομέλεια του Μαρτίου. Boris... Θα... Ο κύριος Μπόρις Γιαροσέβιτς είναι εδώ είναι από την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, από τη σχετική μονάδα. Θέλω να του δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να δηλώσω πω το σχέδιο έκθεση που παρουσιάζεται είναι έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Οι υπηρεσίες μας θα πάνε στην Τασκένδη την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου για τον πρώτο συνολικό γύρο διαπραγματεύσεων για την συμφωνία και οι Ουσμπέκοι έχουν ε, κατεβάσει πολύ εντυπωσιακή ομάδα, το οποίο δείχνει ότι ενδιαφέρονται πραγματικά θα συμμεριστώ τις απόψεις των όσων εδώ μίλησαν και θέλω να τονίσω ένα-δύο σημεία. Καταρχήν η διαδικασία μεταρρυθμίσεων συνεχίζεται. Το 2019 είναι το έτος των ενεργών επενδύσεων και της κοινωνικής ανάπτυξης για το Ουσбекιστάν. Αυτό παρουσιάζει ποιε είναι οι προτεραιότητες. Οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις προχωράνε και για πρώτη φορά οι Standards Poor και οι Fitch του έχουν δώσει ικανοποιητικά, ικανοποιητική βαθμολογία πριν τα Χριστούγεννα ε, στο Σμπέκιστάν. Μιλήσαμε για την πρόσβαση στον ε, ΠΟΕ και θέλει να μπει στη συμφωνία GSP-SYN το Ουσμπεκιστάν και θα πάει και μια αποστολή σχετικά στην Τασκένδη πάλι και αυτή αρχές Φεβρουαρίου. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα Είχαμε την απελευθέρωση των πολιτικών κρατούμενων και θέλω να καταγράψω πως η μεταρρύθμιση στη δικαιοσύνη έδωσε τα πρώτα της αποτελέσματα. Να σας πω πως αυτή τη στιγμή από ε, απελευθερώσεις ε, στο Ουσμπεκιστάν από τις 28 των πολιτικών κρατουμένων πέρσι φτάσαμε τις 600 φέτος. Uh, Έχουμε τη νέα στρατηγική για την ε, Κεντρική Ασία που θα παρουσιάσουμε μέχρι τα μέση Μαΐου και εκεί θα περιγράψουμε ό,τι συμβαίνει στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στο Ουσβέκισταν πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιαρουσέβιτς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα σχόλια. Σας ενημέρωσα για τις ημερομηνίες, για τις τροπολογίες και για την ε, διαδρομή αυτού του θέματος. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο θέμα, το 6. 10 λεπτά έχουμε διαθέσει, που είναι το δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι δυνατότητες για την πρόληψη σειράξεων και για τη διμεσολάβηση. 6 Δεκεμβρίου τα είπαμε για πρώτη φορά. Έχουμε τροπολογίες. Ο κύριος, η κυρία Σοράγια πώς είναι η συγγήτρια και θα της δώσω το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να ξεκινήσω απευθύνονται σε ευχαριστίες μου στους συναδέλφους για ό,τι ε, έδωσαν σε αυτή την έκθεση 182 τροπολογίες πιο συγκεκριμένα οι βασικές ε, αρχές που περιγράφονται είναι η ενίσχυση του θεσμικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη σειράξεων και την διαμεσολάβηση και θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Καταρχήν, η δημιουργία ενός υψηλού επίπεδου ε, συμβουλευτικού οργάνου για την πρόληψη σειράξεων σε συγκεκριμένε χώρες, το οποίο θα ε, ενώσει ε, εμπειρογνώμονες και υψηλά ιστάμενα πρόσωπα από τον πολιτικό κόσμο που θα εξετάζουν τις προτάσεις που υποβάλλει υπό το νέο Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα να ρωτήσω γιατί οι κύριοι Ντανζόν και Καστάλο ζητούν να διαγραφεί αυτή η πρόταση. Δεύτερον, ο διορισμός ειδικού απεσταλμένου για την ειρήνη ε, ή την ε, διαμεσολάβηση και την πρόληψη σειράξεων που ε, επηρεάζουν αμάχους ε, να σας πω πως εδώ φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη μιας ξεκάθαρης εντολής, να το προωθήσουμε σε όλα τα επίπεδα. Ας δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να επισημοποιήσουμε αυτή την εντολή που θα δοθεί. Η δημιουργία επιπλέον διοργανικού ε, μηχανισμού, για παράδειγμα task force, για συγκεκριμένες σειράξεις και την πρόβληψη αυτών, είναι πολύ σημαντική διάσταση και θα βοηθήσει να ενισχύσουμε τις δυνατότητες που έχουμε για την πρόληψη σειράξεων και για τη μεσολόβηση. Είναι ένας οριζόντιος μηχανισμός που είναι πολύ αποτελεσματικός με μια πολύ ρεαλιστική προσέγγιση έτσι ώστε να συντονιζόμαστε και σε επίπεδο ε, κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τόπου. Έχουμε το ομάδα εργασίας του Συμβουλίου ε, η οποία και αυτή είναι απαραίτητη και θα πρέπει το Συμβούλιο ε, να ενισχύσει τη δράση της και να την φέρει στην κορυφή των προτεραιοτήτων. 160 είναι η τροπολογία που θα ήθελα να στηρίξετε, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα δίκτυο διαμεσολαβητών για τις ε, γυναικών ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει κάτι τέτοιο στις βόρειες χώρες και στην Αφρική. Θέλουμε κάτι αντίστοιχο για την Ευρώπη, για την θεσμοθέτηση αυτών των ευρωπαϊκών διαδικασιών. Θα ήθελα να με στηρίξετε στη δημιουργία αυτού του πουλ για που θα είναι πρώην και τρέχοντα μέλη του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης και ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος είναι υπεύθυνο για το συντονισμό αυτών των ε, δραστηριοτήτων. Ο κύριος στάνοκ είπε ότι θα πρέπει να τα συνδέσουμε όλα αυτά στην 163 που ζητά περισσότερο συντονισμό και με τις νομαδεργασίες ε, για τον εκδημοκρατισμό. Θέλω να συμπεριλάβουμε και τις γυναίκες στη διαδικασία ειρήνευσης και θέλω να στηρίξουμε την τροπολογία που στην διαμεσολάβηση και στη διαδικασία πρόληψη σειράξεων θα ενισχύσει το ρόλο τη κοινωνία των πολιτών για τον προπολογισμό. Για να είμαστε αποτελεσματικοί, για να προλαβαίνουμε σειράξει και να μπορούμε να διαμεσολαβήσουμε, θα πρέπει στο επόμενο, στις επόμενες δημοσιονομικές προβλέψεις να έχουμε περιχαρακώσει τα απαραίτητα οικονομικά μέσα προ αυτή την κατεύθυνση. Κάποιοι ζήτησαν το περικαρακώσει του πόρου, ζήτησαν να διαγραφεί και θα ήθελα να μου πείτε γιατί. Επίσης, με χαρά αναμένω τον επικοδομητικό διάλογο που θα γίνει στο πλαίσιο της συνένεσης, του συμβιβασμού και της συνεργασίας. Στη σχετική συνάντηση η οποία θα λάβει χώρα την 5η, 24 του μηνός, σε μια μισή ώρα το μεσημέρι. Θα ψηφίσουμε 2 Φεβρουαρίου στην ΑΦΕΤ για να περάσουμε από την πρώτη ολομέλεια του Μαρτίου. Ευχαριστούμε κύριε Πόστ. Δέκα λεπτά προβλέπονται για τη συζήτηση αυτού του σημείου και έχω έξι συναδέλφους που ζήτησαν τον λόγο. Αλλά έχουμε μείνει 20 λεπτά πίσω. Έχουμε συνολικά 35 σημεία στην ημερήσια διάταξη. 8 80 ε, σελίδες σημειώσει του Πρόεδρου. Νέο ρεκόρ. Οπότε Σα θερμό παρακαλώ να περιοριστείτε στο 1,5 λεπτό. Μίχαλ, εκ μέρου του κ. Ντάνζο, που είναι ο σκιώδη ηγητή του ΕΛΚ, κολλείται δυστυχώ σήμερα, θα διαβάσω τι δηλώσει του. Στόχο του σχεδίου έκθεση είναι να να προτείνει μια σειρά συστάσεων για την ενίσχυση τη ικανότητα Ευρωπαϊκή Ένωση στα θέματα πρόληψη και διαμεσολάβηση τη συγκρούση. Υπάρχουν κάποια θετικά σημεία. Καταρχήν, αντιμετωπίζεται ένα κέριο ζήτημα που βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής διπλωματίας. Η πρόληψη των συγκρούσεων και η διαμεσολάβηση είναι όντως κεντρικά σημεία της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, στόχος να αυξηθεί η ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ ευπρόσδεκτος μέσω της ενίσχυσης των δομών ε, που υπάρχουν στα θεσμικά όργανα για το σκοπό αυτό. Βέβαια, ο κύριος εξακολουθεί να έχει ενδιασμού σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία της έκθεσης. Δεν γνωρίζει πόσο ε, σημαντικέ θα είναι τέτοιου είδου εκθέσει στα τέλη τη θητεία. Και ω προ το περιεχόμενο και την ουσία, και εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα, κατά τη γνώμη του κ. Ντανζάν, γιατί το θέμα τη ε, πρόληψη των συγκρούσεων το εξετάζει μόνο από τη σκοπιά του φύλου, που είναι περιοριστική. Ε, Επίση, το θέμα τη ασφάλεια φαίνεται να αγνοείται πλήρω, να παραμελείται τελείω. Και σίγουρα η ισότητα των φύλων είναι σημαντικό στόχο, αλλά θα πρέπει να είναι ο βασικό σκοπό για την κατάρτιση μια έκθεση. Ο κ. Ντανζάν έχει καταθέσει προτάσει για να εξισορροπηθεί η έκθεση από την άποψη αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γκάλερ. Ο Τσάρλ Τάνοκ από του συντηρητικού μεταρρυθμιστέ. Και εγώ κύριε Πρόεδρε μπορώ με χαρά να συμφωνήσω με μεγάλο τμήμα της έκθεσης. Συμφωνώ πάντως με τον προλαλήσατε ότι θα πρέπει να γίνει κάποια επανισορρόπηση της έκθεσης για να μην επικεντρωνόμαστε αποκλειστικά και μόνο στην προτεραιότητα που δίνουμε στα θέματα ισότητας φύλων. Ε, σημαντικό βέβαια, αλλά υπάρχουν και άλλα σημαντικά θέματα και γι' αυτό έχω καταθέσει σειρά τροπολογιών την 116 ε, για παράδειγμα, την 154. Η 116 μιλάει για την ανάγκη να είναι τελείως, ε, παρόλο που είναι ανεξάρτητο αυτό το θέμα και ιδιότυπο, δεν μπορεί να έχουμε μια ενιαία προσέγγιση για όλα τα ζητήματα. Γιατί το ζήτημα είναι περίπλοκο και οι με μονομένες 154 αφορά μικρή αύξηση των κονδύλων για το βραβείο Ζαχάροφ και ζητώ από τους συναδέλφους ε, να σκεφτούν το γεγονός ότι πάρουμε πολλά κονδύλια για τις ε, αποστολές παρατήρησε εκλογών. Ε, και είχαμε 5.000 ε, για το βραβείο Ζαχάροφ, ε, που είναι πενιχρό ποσό. Μία μικρή στο αύξηση θα ήταν συμβολική αξία για να αναγνωριστεί ο ρόλο αυτών των πρωταθλητών στον ακτιβισμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Και είναι σημαντικό και θεμελιώδη ο ρόλο και η συνεισφορά του στην αποτροπή των συγκρούσεων. Ευχαριστώ. Από την άλλη, κυρία Φόλκμαν. Χωρίς μικρόφωνο δυστυχώς. Δυστυχώς δεν λειτουργεί το μικρόφωνο της ομιλήτριας. Horen jullie mij nu? Ah, oké. Okay. Ja? Now the mic is working. I'm very sorry. Με μικρή καθυστέρηση, ευτυχώς άρχισε και λειτουργεί το μικρόφωνο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την πολύ σημαντική αυτή έκθεση για την πρόληψη των συγκρούσεων και τη διαμεσολάβηση στις συγκρούσεις, βασικά στοιχεία απαραίτητα της εξωτερικής μας πολιτικής. Επίσης, η επένδυση στην προσέγγιση ασφάλεια στις χώρες εταίρους δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των εταίρων μας, αλλά και προς το δικό μας συμφέρον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στα θέματα της πρόληψης και τη διαθέτηση των συγκρούσεων. Και θα πρέπει να προβλέψουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για κάτι τέτοιο και να αναπτύξουμε τις σχετικές μα ικανότητε. Γι' αυτό και στηρίζουμε την έκθεση. Χαίρομαι που δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο ρόλο των γυναικών στην πρόληψη και τη διαμεσολάβηση στις συγκρούσει. Γιατί οι γυναίκε πλήττονται δυσανάλογα από τη συγκρούση, ενώ δεν συμμετέχουν επαρκώ στην αποτροπή ή στη διαμεσολάβηση ε, στι συγκρούσει. Αυτή η κατάσταση θα πρέπει να αλλάξει. Γι' αυτό και έχω καταθέσει πολλέ τροπολογίε που δεν αφορούν μόνο τι γυναίκε, γιατί έχουμε και άλλου ενδιαφερόμενου που θα μπορούσαν επίση να συμβάλλουν στην αποτροπή, η πρόληψη των συγκρούσεων ή στη διαμεσολάβηση. Η νεολαία, για παράδειγμα, είναι, είναι το μέλλον μα. Θα πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στη διαδικασία. Αλλά και άλλοι θα μπορούσαν να λάβουν μέρο σε τέτοιε διαδικασίε. Για να μην ξεχνούμε και ε, στρατιωτικά ε, στρατιωτικούς που επίσης μπορούν να συμβάλλουν στην πρόληψη και διαμεσολάβει της σύγκρουση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Βόλτμανς. Εκπρόσωπος της ΓΚΟΕ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την Σωράγια πόστ για την πολύ αξιόλογη έκθεσή της. Είναι πολύ χρήσιμη αυτή η συζήτηση ε, και για μας για τις τροπολογίες. Οι πράσινοι θεωρούν ότι η διαμεσολάβηση και η πρόληψη συγκρούσεων είναι σημαντικό καθήκον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι, αν τι άλλο παράδοξο, να αφιερώνουμε μόνο ένα δεκάλεπτο για μια τόσο σοβαρή έκθεση και ένα τόσο μείζον ζήτημα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εμβαθύνει σε αυτή τη συζήτηση με πολυτέλεια χρόνου. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε δυστυχώ λίγο χρόνο στη διάθεσή μα, γι' αυτό και καλό θα ήταν να επικεντρωθούμε στα απολύτω απαραίτητα. Για παράδειγμα, στο μακροπρόθεσμο προπολογισμό, στην ανάγκη ενίσχυση ε, τη πολιτική εξουσία ε, και τη σχέση μα σε ό,τι αφορά θέματα πρόληψη συγκρούσεων και διαμεσολάβηση τη συγκρούση. Σίγουρα το, ο μηχανισμός για τη σταθερότητα και την ειρήνη που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ουσιαστικά ακολουθεί μια πολιτική λιτότητας. Σφίγγουμε συνέχεια το ζωνάρι. Αναφέρθηκαν τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας και για, την, για τους εξοπλισμούς στρατιωτικούς και για την ενίσχυση του στρατιωτικού σκέλους των δράσεών μας, αλλά γιατί δεν επενδύουμε και στο πολιτικό σκέλος. Εδώ δεν έχουμε ούτε 3 δισεκατομμύρια και κονδύλια που δεν θέλετε να είναι ειδικού σκοπού και προσημειωμένα για συγκεκριμένο στόχο. Και ίσως αυτός ο μηχανισμός σταθερότητας και ειρήνης τελικά ε, εξαφανιστεί λόγω του πενιχρού προπολογισμού που προβλέπετε. Πιστεύω ότι χρειάζεται πιο στενή συνεργασία για τα θέματα αυτά. Θα καταθέσω και τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Βαλέρο. Ο κύριος Κόουσο. Για μας, οποιαδήποτε πρωτοβουλία που έχει σκοπό να προωθήσει μηχανισμούς για την πρόληψη και την μεσολάβηση σε σειράξεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλοδεχούμενη. Αλλά αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από την καλή πρόθεση ε, και οι μηχανισμοί αυτοί να επιτηρούνται και να ελέγχονται με δημοκρατικό τρόπο. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν θα πρέπει να αποτελούν απλή δήλωση καλών προθέσεων, αλλά θα πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις έτσι ώστε οποιαδήποτε τέτοια πρόταση να είναι αποτελεσματική. Εκτιμάμε πολύ θετικά αυτή την ολοκληρωμένη απόκριση που θα δίνουμε στην πρόληψη σειράξεων, όπως επίσης και στον ειδικό απεσταλμένο για την ειρήνη και άλλους διοργανικούς μηχανισμούς. Είναι σημαντικό το σημείο 11 για μας, πρόσβαση στις πληροφορίες και πιο συγκεκριμένα με ένα φόρματ που θα το κάνει εύκολο. Αυτό είναι ζωτική σημασία για την πρόληψη και τη διαμεσολάβηση. Ο μηχανισμός αυτός θα πρέπει όμως να έχει ένα ρόλο σημαντικό συνεργαζόμενος πάντα με διεθνείς οργανισμούς και κυρίως τον ΙΟΙΕ και τις υπηρεσίες του. Και αυτή θα είναι η δική μας πρόταση. Ευχαριστώ. Thank σας ευχαριστώ κύριε Κόσου. Δεν υπάρχουν άλλα, άλλα σχόλια από τη δική σας πλευρά, οπότε θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Ξέρετε, 4 Φεβρουαρίου στην Επιτροπή μας θα ψηφίσουμε και ελπίζω να τα καταφέρουμε με, για την Ολομέλεια 11 με 14 Μαρτίου. Στο επόμενο σημείο, που είναι το 7, εκλογές στη Γεωργία 20 Οκτωβρίου και 20 Νοεμβρίου και πέρσι επίσης τις πρόορες εκλογές στην Αρμενία, τις βουλευτικές στις 9 Δεκεμβρίου και στις δύο χώρες και στις δύο περιπτώσεις στείλαμε 6 με 7 μέλη ε, του Κοινοβουλίου ως ε, παρατηρητές, εκπροσωπούν τις περισσότερες από τις ομάδες. Ο κ. Κίνε ήταν ε, για τη Γεωργία και ήταν η Χάουτι Χάουτ, αλλά που στην Αρμενία. Εμείς συνεργαστήκαμε όπως πάντα στα πλαίσια του, της αποστολής του ΟΑΣΕ ε, και στη Γεωργία μαζί με τον ΝΑΤΟ, στην Αρμενία και στη Γεωργία επίσης με το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Θέλω και οι δύο που ηγήθηκαν αυτών των αποστολών, αλλά και τα υπόλοιπα μέλη, να μα κάνουν ένα debriefing. Μου είπατε, μου είπαν μόνο ε, ο Ιωαχέμ Τσέλερ είναι ο πρώτο που θα λάβει το λόγο για να αντικαταστήσει τον συνάδελφό του. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Αντρική. Ε, δεν θα μπορούσε να έρθει δυστυχώς ε, ασθενή. Και έτσι ερχόμενος εδώ στην Βρυξέλλες έλαβα το μήνυμα ότι με παρακαλεί να αναλάβω, να σας ενημερώσω για τις προεδρικές εκλογές στην Γεωργία. Όπως είπατε και εσείς, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έστειλε έξι μέλη ως παρατηρητές ε, στον πρώτο γύρο της, της προεδρικής εκλογικής αναμέτρησης. Δύο είναι Στο, εφόσον στον πρώτο δεν εξασφάλισε κανένας από τους υποψηφίους την απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται μια δεύτερη ψηφοφορία. Και ως ήθεστε κράτη του όπως γίνεται και με τα άλλα κράτη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητήθηκε από την ε, ΟΑΣΕ να αναλάβει τις, ε, ε, την παρατήρηση των εκλογών. Είχαμε και άλλες αποστολές κοινοβουλευτικών παρατηρητών από κοινοβουλευτικές συνελεύσεις. Στο πλαίσιο των διεθνών αποστολών παρατήρησης, συντονιστής ο Κρίστιαν Βίτζενιν, πρώην συνάδελφος και τώρα βουλευτής στο Βουλγαρικό Κοινοβούλιο. Είχαμε εκπροσώπους από την ε, Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΟΑΣΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και του ΝΑΤΟ. Το πρόγραμμα το είχε ετοιμάσει ο ΑΣΕ για όλους τους βουλευτές και πρόβλεπε συναντήσεις με τους ε, πιο προβεβλημένους υποψηφίους κτλ. Πέραν αυτών, η αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου είχε και την ευκαιρία να συναντηθεί με τον περχόμενο πρόεδρο, τον, Υπουργό, ε, τον Πρωθυπουργό συγγνώμη, Μπαχτάτσε και με προσώπους των πρεσβειών των κρατών μελών αλλά και με τον επικεφαλής της ε, εκεί αντιπροσωπείας μας. Όπως είπα, στον πρώτο γύρο από τους 25 υποψηφίους κανένας δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία. Έτσι λοιπόν στις 28 Νοεμβρίου έλαβε χώρα ο δεύτερος γύρος, ο πρώτος ήταν στις 28 ε, Οκτωβρίου. Με το δεύτερο αυτό γύρο λοιπόν έγινε η τελική αναμέτρηση μεταξύ της ε, Σάλομε Σουραμπισβίλη που κατέβηκε ως ανεξάρτητη υποψήφιος, αλλά ήταν προφανές πως ε, στην πραγματικότητα τη στήριζε το κυβερνών κόμμα και κέρδισε τις εκλογές με το 59,5% των ψήφων, ενώ ο αντίπαλος από το κόμμα UNM, Γκριγόρ Βαλσάτσε, κέρδισε το 45% περίπου των ψήφων. Στον πρώτο γύρο ήταν πολύ κοντά οι δύο υποψήφοι, είχαν ένα 37-38% ο καθένας. Η Σάλομε Ζουραβισβήρη λοιπόν αναλαμβάνει καθήκοντα στις 16 Δεκεμβρίου του 2018 ω πρόεδρος της Γεωργίας και ορκίζεται. Ήταν ε, η τελευταία φορά που εκλογική, η προεδρική εκλογή έλαβε χώρα με άμεση ψηφοφορία καθώς ύστερα από αναθεώρηση του συντάγματος ε, από εδώ και μπρος θα είναι έμεση από το κοινοβούλιο, δηλαδή θα αναδεικνύεται ο πρόεδρος. Η... Ο κύριος Ανδρικένε μου έχει δώσει τα στοιχεία αυτά που ήθελε να σας διαβάσω στα αγγλικά. Και είναι εξή πολλά μπορούμε να πούμε για τις εκλογές και τη διαδικασία αυτή καθεαυτή. Αναφερόμαστε καταρχάς στη, στην ε, διαδικασία την ίδια. Ήταν επαγγελματικός ο τρόπος διεξαγωγής των εκλογών. Η προεκλογική εκστρατεία ήταν ελεύθερη και οι προσβασίες στις κάλπες επίσης δεν υπήρξαν την ημέρα των εκλογών παρά κάποιους φόβους έκτροπα. Μεταξύ των δύο γύρων υπήρχε μια ομαλότητα, αν και πρέπει να πούμε ότι στον πρώτο γύρο ήταν στο 50% και χαμηλότερη προσέλευση. Ίσως θα περιμέναμε περισσότερο ενδιαφέρον από τον ψηφοφορό και συνεχίζω με το κείμενο του συναδέλφου. Δυστυχώς κάποια στοιχεία αμάβρωσαν την, διαδικασία, την εκλογική διαδικασία. Αρχικά υπήρξε πολύ αρνητική εκστρατεία και προπαγάνδα με πολύ σκληρές κατηγορίες ε, εις βάρος των αντιπάλων με πολύ ζωφέρες εικόνες που αναφέρονταν στο μέλλον της χώρας. που διωγγώθηκαν ιδιαίτερως μετά και στο δεύτερο γύρο, ενώ του δεύτερου γύρου, όπως άλλωστε σημειώθηκε στο δεύτερο γύρο επίσης ε, παρουσιάστηκε μεγαλύτερη πόλωση στον τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που δεν εξασφάλισαν ισότιμη πλατφόρμα παρουσίασης. Οι ανεξάρτητες οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών κατέστησαν στόχοι επιθέσεων στοχευμένων από διάφορες πλευρές αλλά και απειλών. Καταδικάστηκε αυτό από το, την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στον πρώτο γύρο και αυτό φαίνεται να επίδρασε θετικά γιατί φάνηκε, φαίνεται πως ε, στο δεύτερο γύρο τέτοιου είδους φαινόμενα να ήταν λιγότερο έντονα. Πάντω βλέπουμε βελτίωση σε σχέση με τις εκλογές του 2016, ε, ανισορροπία σε σχέση με τους πόρους. Βλέπουμε ότι είχε πολύ περισσότερες δωρεές η λέξη το κυβερνών κόμμα σε σχέση με όλους τους άλλους, ο υποψήφιο του κυβερνώντο κόμματο, η υποψηφία του κυβερνών κόμματο σε σχέση με όλους τους άλλους. Ε, υποψηφίους συνολικά. Υπήρξαν ζητήματα διασπάθησης ε, κονδυλίων, ε, όπως η με την ανακοίνωση μερικές μέρες πριν από το δεύτερο γύρο της αποπληρωμής των προσωπικών δανείων περί των 600.000 πολιτών, δηλαδή περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ από αρχές, από το κυβερνών κόμμα, εν περιπτώσει. Κατά την ημέρα των εκλογών υπήρξαν κάποιες ενδείξεις για εκφοβισμό, απειλές από εκπροσώπους εντό εισαγωγικών των κομμάτων που ήταν ε, παρόντες στα εκλογικά τμήματα και ε, μαζικής εκστρατείας μέσω σύντομων μηνυμάτων τηλεφωνικών ή και τηλεφωνημάτων ακόμη, παρότι αυτό δεν απαγορεύεται από τον νόμο. εν όλο και παρά κάποιες θετικές εξελίξεις, ο δεύτερος γύρος φαίνεται να δίνει χειρότερη εικόνα από ότι ο πρώτος. Πολύ μεγαλύτερη δηλαδή ήταν η πόλωση στην κοινωνία και αυτό θα απαιτήσει μεγαλύτερη διαδικασία για αποκατάσταση των πληγών. Οι ε, παρατηρήσεις και οι επικρίσεις του Κοινοβουλίου και για τους δύο γύρους ήταν σαφείς και έντονες περιμένουμε για τη χώρα αυτή που έχει και πρώτη θέση στην περιοχή να προχωρήσει προς τον δρόμο της δημοκρατίας. Τα αρνητικά στοιχεία είναι σημαντικό να μην επικρατήσουν, να μην παγιωθούν ως τάση, δεδομένου δε ότι υπάρχουν και εκλογές το 2020 για το Κοινοβούλιο, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η τήρηση των ε, συστάσεων από τις αρμόδιες αρχές και η ε, προσαρμογή στις πολιτικές ε, εξελίξεις στη γεωργία ε, βεβαίως θα πρέπει να συνδυαστούν και με την επίλυση των ζητημάτων των καταχωμένων εδαφών. Ευχαριστώ πολύ, Γιωάχιμ Τσέλερη. Τώρα η κυρία Χάουταλα, που μόλι. έφτασε. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά θα σας ενημερώσω για την αποστολή παρατήρηση εκλογών στις πρόορες ε, βουλευτικές εκλογές που έγινε στην Αρμενία στις 9 Δεκεμβρίου ε, του προηγούμενου έτους και μάλιστα σε ένα και μόνο γύρο. Όπως πάντα είχαμε μια άρτια αντιπροσωπή εξαμελή για την παρατήρηση εκλογών, τέσσερις υπαλλήλου και οι ευρωβουλευτές ήταν Φαρία, Πιτέλα, Πιτέρα, ε, Φίσας, ε, Μούντι και Χάρμς και υποφαινόμενοι φυσικά. Και μάλιστα ε, φτάσαμε στο Γερεβάν τρεις μέρες πριν την διεξαγωγή των εκλογών και ενημερωθήκαμε εκτενώς από το ΝΤΙΡ, την, μακρο... την αποστολή μας και από ενδιαφερόμενους εκπροσώπους των κομμάτων, κοινωνία των πολιτών και μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ε, στις σαφές ε, σε αυτές τις σημαντικές συναντήσεις που είχαμε ότι οι τελευταίες εκλογές ήταν πολύ διαφορετικές από όλες τις προηγούμενες εκλογές της Αρμενίας πριν τις εκλογές πριν την Επανάσταση που έλαβε χώρα στο Απρίλιο και Μάιο του 2018. Και στα συμπεράσματα που συντάξαμε με τους συναδέλφους από το Συμβούλιο της Ευρώπη και την ΟΑΣΕ και τα οποία προσυπογράφουμε πλήρως, τονίσαμε ότι οι συγκεκριμένε εκλογές έγιναν με σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών με, ε, και με τη λαϊκή εμπιστοσύνη που θα πρέπει να διαφυλαχθεί και στι επόμενε εκλογικέ μεταρρυθμίσει. Επίσης ε, και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, συνέβαλα σε μια σημαντική εκστρατεία παρόλο που υπήρχε κάποια ε, ρητορική στο έντονη ρητορική στο διαδίκτυο κυρίως. Κάτι που, να, ε, που ήταν σημαντικό πρόβλημα και σε εκλογές του 2017. Γενικώ ε, καταλήξαμε στην, ε, στα κρούσματα ακόμη και χρηματισμού των κάποιων ψηφοφόρων. Αυτή τη φορά όμως δεν ε, υπήρχαν τέτοια φαινόμενα και ήταν πραγματικά θεμητός ανταγωνισμός μεταξύ των κομμάτων και οι εκλογές έγιναν ήρεμα ε, και αξιολογήθηκαν πολύ θετικά και μάλιστα ήταν πρόορες αυτές οι εκλογές και πολύ γρήγορε. Υπήρχε λίγο χρόνος για την προεκλογική εκστρατεία, γιατί έγιναν σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Πάντως ήταν αξιοθαύμαστο πόσο αποτελεσματικά η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή κατάφερε να διοργανώσει τη διαδικασία Πρόσκοπτα και να ε, γίνει σωστή εφαρμογή του εκλογικού νόμου. Αναγνωρίζουμε λοιπόν τη σημαντική αυτή, το σημαντικό αυτό επίτευγμα της Κεντρικής ε, Εκλογικής Επιτροπής σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Κάποιες ε, επικριτικές παρατηρήσεις αφορούσαν περισσότερο το νομοθετικό πλαίσιο παρατηρήσαμε για παράδειγμα κάποια προβληματικά σημεία με τη χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας, τη, τις απαιτήσει ε, για την ηθαγένεια, τους καταλόγους ε, ψηφοφόρων και την ανάγκη της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική διαδικασία. Αυτά τα σημεία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεταρρυθμίσεις στην νομοθεσία και προσβλέπουμε σε άμεσες τέτοιες εκλογικές μεταρρυθμίσεις. Και ελπίζω αυτό να εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα και της ε, Βουλής Αρμενίας και της αρμενικής κυβέρνησης. Θα πρέπει οποιαδήποτε μεταρρύθμιση να γίνει με συμμετοχή και της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών και όλων των ενδιαφερομένων μερών. Επίσης, ε, ήταν συμμετοχή, ε, έντονη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην εκλογική διαδικασία. Βέβαια, πραγματικά ήταν εξωθαύμαστη αυτή η συμμετοχή και ήταν πολύ ενθαρρυντικό που για πρώτη φορά ακούσαμε τόσο πολλούς εκπροσώπους κοινωνίας των πολιτών να συμφωνούν με εκπροσώπους και των πολιτικών αρχών και των κομμάτων για τον τρόπο διεξαγωγή των εκλογών. Κάτι που εξασφάλισε σημαντική εμπιστοσύνη του κοινού, του λαού στην εκλογική διαδικασία. Και μετά την λήψη του 70% των ψήφων για το κόμμα του και Πρόεδρου Μπασίνιαν, υπάρχουν υψηλές προσδοκίες για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και τη βελτίωση των βιωτικών συνθήκων στην Αρμενία. Τους τελευταίους μήνες όπως ξέρετε, η Αρμενία, βρέθηκε στη, στο πρόγραμμα της εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ό,τι αφορά τις διμερείς σχέσεις, υπογράψαμε και εφαρμόζουμε προσωρινά την ε, ε, ενισχυμένη εταιρική σχέση, που θα αποτελέσει και το δοδικό χάρτη συνεργασίας με σημαντικέ μεταρρυθμίσει και χρηματοοικονομική ενίσχυση. Και αν η αρμενική κυβέρνηση ζητήσει περαιτέρω ε, υποστήριξη για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων, των μεταρρυθμίσεων, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να την επικουρήσουμε. Και αυτό ευθυγραμμίζεται με τι δεσμεύσει μα για την εμβάθυνση των σχέσεών μα με την Αρμενία, κάτι που είναι προ όφελο όλων των πολιτών τη χώρα αυτή. Θα ήθελα τέλο να ευχαριστήσω θερμότατα του συναδέλφου ευρωβουλευτέ, του συναδέλφου από τι άλλε κοινοβουλευτικέ συνελεύσει και κυρίω τον πρέσβη Ζουλαγκάσεκ και το επιτελείο του για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε επί τόπου. Επίση, θα ήθελα να ευχαριστήσω το πρέσβη Πιόταρ Σβιτάρσκι και την ομάδα του για την βοήθεια που μας έδωσε στη διάρκεια της αποστολής. Μπορούμε λοιπόν στην περίπτωση αυτή να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η έκβαση όντως ήταν αντανάκλαση της ε, λαϊκής βούλησης, κάτι που δεν ίσχυε για τις προηγούμενες εκλογές του Απριλίου του 2017. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Χάουταλα για την ενημέρωση. Και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Σατζίτ Καρίμ, που είναι η Δήμον για την ευρύτερη περιοχή. Από Σας καλωσορίζουμε και στην Επιτροπή ΕΦΕΤ. Σας ευχαριστώ. Ήσασταν πάρα πολύ γενικό στην εισαγωγή, οπότε ακόμα και εγώ περιμένω με αγωνία να ακούσω τι θα πω. Εν πάση περιπτώσει θα ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους τους συναδέλφους οι οποίοι ανέλαβαν να ταξιδέψουν εκ μέρους ε, ολόκληρου του Κοινοβουλίου. Ξέρω πως η Χάιντι το έχει ξανακάνει και έχει ξαναπάει σε τέτοιου είδους αποστολή στην Αρμενία και το γεγονός πως συμμετείχαμε κι εμείς ως ε, όργανος σε αυτό το σώμα ε, παρατηρητών ήταν πάρα πολύ σημαντικό και στην περίπτωση Γεωργίας και στην περίπτωση Αρμενίας στις εκλογές στην Αρμενία που έγιναν 9 Δεκεμβρίου, όπως είπε η Χάιντι, ήταν ε, προώρες εκλογές και η γενικότερη άποψη από τη δική μας ε, αποστολή, αλλά γενικότερα, Η άποψη λοιπόν είναι πως αυτές οι εκλογές σεβάστηκαν τις θεμελιώδεις ελευθερίες και στηρίχθηκαν ευρύτερα από το κοινό και αυτές τις ε, κακές πρακτικές που είχαμε δει στο προηγούμενο σε άλλες εκλογές της Αρμενίας δεν τις ξαναείδαν οι παρατηρητές μας. Και επειδή είμαι ο πρόεδρος της αντιπροσωπείας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον Νότιο Κάυκασο, εντυπωσιάζομαι από την πρόοδο που έχει κάνει η Αρμενία τους τελευταίους μήνες. Μετά την Βελούδινη Επανάσταση, οι εκλογές αυτές δεν ήταν μόνο ε, ένα οριακό σημείο για τη δημοκρατία στη χώρα αυτή, αλλά και ένα, μια μεγάλη δοκιμασία και για τη νέα κυβέρνηση, αλλά και για την εμβάθυνση των νέων σχέσεων που έχουμε ε, με τη χώρα αυτή. Για τον Νικόλ Μεσανιά να σας πω πως ήρθε σε συνάντηση πολλές φορές με τη δική μας αντιπροσωπεία για τον Νότιο Κάυκασο και πριν γίνει πρωθυπουργό και τώρα και νομίζω ότι και εσείς Πρόεδρε είχατε ε, πάει μια φορά σε μια αποστολή που στείλαμε και είχατε συναντηθεί και εσείς μαζί τους και οι ελπίδες μας ήταν ε, η εντολή του να ενισχυθεί ε, σε σχέση με το παρελθόν και να νομιμοποιείται και φαίνεται πως σήμερα είμαστε στη θέση να το πούμε αυτό. Έτσι λοιπόν έχω την πίστη πως η Αρμενία θα είναι ψηλά στο θεματολόγιο με τις προτεραιότητες εξωτερικής πολιτικής της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να επικυρωθεί η συνθήκη με όλα τα κράτη-μέλη από όλα τα κράτη-μέλη και αυτό προς όφελος και των Ευρωπαίων πολιτών αλλά και της Αρμενίας. Η επόμενη συνάντηση της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής θα γίνει το φθινόπωρο και εκεί θα κάνουμε και μία απογραφή της προόδου που θα έχει σημειωθεί στο θέμα αυτό. Τέλος, για τη Γεωργία, να σας πω πως άκουσα τα όσα είπε ο συνάδελφος για την ε, αντιπροσωπεία εκεί. Να σας πω πως η Γεωργία τα τελευταία δέκα χρόνια έχει κάνει πάρα πολλές προσπάθειες εδώ και πολλά χρόνια να ενισχύσει τη φήμη της ε, ως πρωταγωνιστή και πρωταθλητή σε επίπεδο δημοκρατίας και εκδημοκρατισμού στην περιοχή εκείνη. Βέβαια, στη συγκεκριμένη εκστρατεία είχαμε πολύ αρνητική προεκλογική εκστρατεία από πολλούς, με πολύ έντονες επιθέσεις κατά της κοινωνίας των πολιτών από τις αρχές, κάτι το οποίο εμείς τονίσαμε. Και βέβαια είχαμε και τα διάφορα επεισόδια, ε, τα γνωστά, που δεν θα έλεγα πως αποτελούν μια γενικότερη τάση και τα οποία δεν θα πρέπει να μας ε, παρασύρουν από το να πιστέψουμε πως είχαν τη δυνατότητα να κάνουν ελεύθερη προεκλογική εκστρατεία ή υποψήφια. Κάτι που με ανησυχούσε εμένα ιδιαίτερα. Η επόμενη συνάντησή μας θα γίνει 28 Μαρτίου και ενδεχομένως ίσως είναι και το τελευταίο που θα κάνω επισήμως ως Ευρωβουλευτής. Το Brexit ξεκινά 29 Μαρτίου, ζούμε λοιπόν εκεί τι θα γίνει. Πάντως εγώ θα κάνω ό,τι μπορώ στα θέματα αυτά. Να θίξω ότι υπάρχει και με τους ομολόγους μας και με την καινούρια ε, Προέδρου, την Σαλόμη Ζουραμπασβίλη που θα επισκεφτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα είναι μάλιστα εδώ αύριο. Και θεωρώ πως η εκλογή της αν δούμε πέραν των ε, πρακτικών που συνδυάζονται με τις εκλογές, είναι ένα πολύ καλοδεχούμενο γεγονός. γυναίκα πρόεδρος στη Γεωργία, αυτό λέει πάρα πολλά. Και είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία ε, και πιστεύω πως τη θέση που έχει αναλάβει θα βοηθήσει στο να εμβαθύνουμε και να ενισχύσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις. Και ελπίζω πως αυτή την, σε αυτή τη θητεία της θα προσπαθήσει να συμφιλιώσει τη χώρα γιατί είναι πάρα πολύ πολλωμένη και κοιτώντας και την Ευρώπη πιστεύω πως όλοι έχουμε τέτοια θέματα πόλωσης και οι δυνάμεις που θέλουν την πόλωση ενισχύονται παντού. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να επενδύσουμε στο να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με τη γεωργία και να προσφέρουμε και την απαραίτητη και βοήθεια σε κάθε περίπτωση όπου μπορούμε. Σας ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ πολύ. Τρεις συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Γκόμες, Μούντι, Χάρμς. Δύο λεπτά εκάστε, κύριε Γκόμες, πρώτα. Ναι, συμφωνώ απολύτως ε, στα όσα είπε από την ανακοίνωση ο κύριος Τσέλερ που μας τη διάβασε και είναι ευπρόσδεκτες βεβαίως ε, οι προτάσεις και των συναδέλφων. Ε, βεβαίως ήταν, υπήρχε ανταγωνισμός στις εκλογές αυτές και πάνω απ' όλα σε σχέση με τις ε, κοινοβουλευτικές εκλογές του 2016 δεν υπήρχε βία. Τότε είχα ηγηθεί εγώ της αντιπροσωπείας μας. Πιο δύσκολο να δεχθεί κανείς ήταν αυτό το θέμα της πόλωσης και το πώς ε, είδαμε να εξελίσσεται και σε ορολογία ακόμη δεδομένου ότι η υποψήφια ήταν η γυναίκα, ε, πολύ δυσάρεστη. Αλλά και οι επιθέσεις κατά τις των μη κυβερνητικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που περιέγραψε και ο κύριος Τσέλερ. Μας προβλημάτισε επίσης ιδιαίτερος η παρέμβαση στο συγκεκριμένο επίπεδο βεβαίως, γιατί θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα. και τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, δηλαδή αμέσως πριν από το δεύτερο γύρο. Γιατί δεν μπορεί να είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια για παρέμβαση. Και οι δεσμοί με τον ολιγάρχη αυτόν από την τράπεζα που χρηματοδοτούσε τα δάνεια και το κράτος, τις κρατικές αρχές, δεν μας αφήνει παρά μια δυσάρεστη γεύση. Πάντως οι Γεωργιανοί είναι έξυπνοι άνθρωποι. Παρά τα συνηθισμένα, η απαράτσιξη είναι πάντοτε στα εκλογικά κέντρα, ελέγχουν κτλ. Ο, ο κόσμος είναι έξυπνος και έχει καταλάβει και το βλέπουμε και στα αποτελέσματα του πρώτου γύρου. Και στο δεύτερο γύρο μπορώ να πω ότι πάλι η ξυπνάδα δείξανε επιλέγοντας ε, το αποτέλεσμα το οποίο δεν θα έφερνε την ε, καταστροφή, γιατί ξέρουν ότι ένα άλλο αποτέλεσμα θα έφερνε μια καταστροφή, θα πολύ δυσάρεστη ατμόσφαιρα. Και γι' αυτό ελπίζω να μπορέσουμε για τις προσεχείς γενικές εκλογές το 2020 να αποφύγουμε την πόλωση. Ευχαριστώ. Κυρία Μούντι για την ε, γεωργία. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίζεται η έκβαση της έκθεσης και να υπογραμμίσετε ότι ήταν ε, καθαρή η επιλογή του λαού. και σε σχέση με την ταξινόμηση στην ε, Δημοκρατία και τα Δικαιώματα. Είδαμε ότι η Γεωργία το 2018 είχε, κατα... Ναι, είχε καταχωρηθεί ως, ε, σε μια θέση υψηλότερη από τρεις δικές μας ευρωπαϊκές χώρες. Αισιόδοξο επίση μήνυμα αποστέλει η επιλογή γυναίκας Προέδρου, όταν έχουμε λιγότερο από 10% των γυναικών στο παγκόσμιο επίπεδο σε τόσο υψηλά αξιώματα και παρά τις επιθέσεις που δέχτηκε. Γιατί το βλέπουμε και αυτό. Όταν οι γυναίκες κατεβαίνουν ε, υποψήφιες, ε, πέφτουν θύματα στοχευμένων προσωπικών επιθέσεων. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να γνωρίσουμε ότι την ε, γυναίκα υποψήφια για πρόεδρο που ήταν και πολύ ικανή ιδιαίτερα για το ρόλο των εξωτερικών, της εξωτερικής εκπροσώπης που είναι κατά κύριο λόγο ο ρόλος ε, του Προέδρου της Γεωργίας, της Προέδρου της Γεωργίας, την υποστήριξαν 60% των ψηφοφόρων περίπου. Για την Αρμενία. Είχα τη χαρά να συμμετάσχω στην αποστολή παρακτήρησης και ευχαριστώ τη Χάιντι για την εξαιρετική καθοδήγηση των εργασιών μας. Και πάλι βλέπουμε μια μετάλλαξη στην εκλογική διαδικασία στην Αρμενία. Πριν από έξι μήνες, μέσα σε έξι μήνες μάλλον δεν μπόρεσε να αλλάξει ο εκλογικός νόμος, αλλά ελπίζω αυτό να συμβεί στο μέλλον. Περιμένω το δω και βεβαίω προσβλέπω και στι επιτυχεί εκλογικές αναμέτρησεις. Ευχαριστώ, η Ρεμπέκα Χάρμ. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η περίοδος ε, για τις χώρες ανατολικής γειτονία. Μετά τις εκλογές στη Γεωργία και την Αρμενία, πολύ σύντομα θα έχουμε εκλογές και στη Μολδαβία και στην Ουκρανία. Και μάλιστα στην Ουκρανία δύο φορές θα έχουμε εκλογές ε, για τις προεδρικές εκλογές και τις βουλευτικές και μετά τα πρώτα εκλογικά αποτελέσματα και τις εκλογές στη Γεωργία και Αρμενία, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν αρκετά κοινά σημεία, κάποιες ομοιότητες μεταξύ των ε, εταίρων της Ανατολικής Γειτονίας, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και σημαντικές διαφορές και διαφορετικές εξελίξεις. Ε, και αυτό χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και φυσικά σημαντική δέσμευση. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Με κάλυψε πλήρω η Χάιντι για την Αρμενία. Ήταν πραγματικά μια πολύ καλή στιγμή για μας, ε, για την παρουσία των Ευρωπαίων εκεί. Και ακούσαμε τόσο πολλούς ε, και διαφορετικούς συνομιλητές που μας εξήγησαν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της Αρμενίας θα έχουν πραγματικά ελεύθερες εκλογές ε, και πολλοί μας είπαν ότι αυτή η κατάσταση είναι προηγουμένου γιατί για πρώτη φορά δεν γνώριζαν πριν τις εκλογές το αποτέλεσμα. Και τώρα που σχηματίζεται η νέα κυβέρνηση, οι προκλήσεις είναι πολλές. Και φυσικά πολλές οι προσδοκίες που έχει γύρει ο νέος Πρωθυπουργό, γιατί δεν θα πρέπει μόνο να αξιολογηθεί η θετική διαδικασία των εκλογών, αλλά θα πρέπει τώρα να περάσουμε στη φάση της εφαρμογής της συμφωνίας και να στηρίξουμε τη νέα κυβέρνηση που βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωστρατηγική κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τη Γεωργία απογοητευθήκαμε αρκετά. Παρά το γεγονό ότι έχουμε για πρώτη φορά γυναίκα πρόεδρο, αυτό το αποτελέσμα με ικανοποιεί μεν, αλλά ε, μείναμε απογοητευμένοι από την όλη διαδικασία. Πάντως ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την αυριανή επίσκεψη της συνεκλογής σας Πρόεδρου για να συζητήσουμε με, με τους φίλους της Γεωργίας και όλους όσους στηρίξαμε τη Γεωργία τα τελευταία χρόνια να δούμε πώς θα την ενθαρρύνουμε για να ακολουθήσει αυτό το θετικό δρόμο και πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε κυρία Χάρμς. Δεν ζήτησε άλλο κανεί το λόγο, οπότε να σας να δώσω το λόγο στο Ρίτσαρτ για σύντομα σχόλια. Ευχαριστώ και χαίρομαι και εγώ που έρχομαι για πρώτη φορά εδώ από τότε που ανέλαβα καθήκοντα τον Οκτώβριο. Οι εκλογές στη Γεωργία ήταν πολύ σημαντικές. Ήταν οι τελευταίες ε, προεδρικές εκλογές με άμεση ε, εκλογή και ήταν ένα, μια δοκιμή διάμεση για την κυβέρνηση. Και μάλιστα η πλειοψηφία ήταν 60% για τον πρόεδρο. Δεν θα επαναλάβω τις παρατηρήσεις που μας έκαναν τα μέλη της, της αποστολής παρατηρήσεις εκλογών. Υπήρξε αρκετό ανταγωνισμό αυτό το θετικό, αλλά το αρνητικό ήταν ότι έγινε κατάχρηση των διοικητικών κονδυλίων, υπήρξαν ανισορροπίες στη χρηματοδότηση των κομμάτων και αρκετή πόλωση στη δημόσια συζήτηση και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πάντως θα χρησιμοποιήσουμε τώρα το πολιτικό διάλογο που έχουμε με τη Γεωργία για να, τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπιστούν αυτές οι ελλείψεις και δυναμίες και οι στάσεις του ΟΝΤΙΡ είναι πολύ σημαντικές εν ώψη των ε, βουλευτικών εκλογών που θα γίνουν του χρόνου. Ο, πάντως η πρόεδρος ε, Γιώργος Βίλης στην ομιλία της ε, τόνισε την την ευρωπαϊκή προοπτική της γεωργίας και τον προσανατολισμό της και την πρόθεσή της να ξεπεραστεί η πόλωση αυτός ο διχασμός ε, της γεωργίας και να είναι πρόεδρος όλων των Γεωργιανών Πολιτών. Θα συναντήσει αυτή τη βδομάδα στην Βρυξέλλες τους πρόεδρους Τούσκ Ταγιάννη, καθώ και την είπατε εκπρόσωπο Μογγενή και τον κύριο Αβραμόπουλο. Πολύ σημαντική ευκαιρία λοιπόν για να ξεκινήσει ο διάλογο με τη νέα πρόεδρο, να δούμε τι προτεραιότητες κατά την εξαίρετη θητεία τη και γιατί στο η συνταγματική αναθεώρηση περιορίζει τους προεδρικές εξουσίες. όλα αυτά θα είναι σημαντικός εκπρόσωπος της Γεωργίας ο πρόεδρος στη παγκόσμια σκηνή και χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την πρώτη γυναίκα πρόεδρο στη Γεωργία. Πάντως θα λάβουμε υπόψη τη σημασία που έχει η πολυφωνία, ο πλουραλισμό στη Γεωργία και η επανασυμφιλίωση, η ανάγκη υλοποίηση και ολοκλήρωση μάλλον της συνταγματική αναθεώρησης και να δούμε το νέο εκλογικό νόμο και το νέο σύστημα που θα τεθεί σε ισχύ στο μέλλον. Πάντως αυτά για τη Γεωργία και την Αρμένη είχαμε πολύ σημαντικέ εκλογές που ολοκλήρωσαν την περσινή επανάσταση και το κόμμα My Step του κ. Πασινιάν το βήμα μου συγκέντρωσε την ε, μεγάλη πλειοψηφία στη Βουλή σε σχέση με το Ριπομπλικανικό Κόμμα που δεν ε, μπόρεσε καν να συγκεντρώσει το κατόφλι του 5% για να μπει στη Βουλή. Οι ευρωβουλευτές μίλησαν για το σημαντικό ρόλο που άσκησε η κοινωνία των πολιτών και η εκλογική ε, αρρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση των εξοπλισμών των εκλογικών κέντρων και στην ε, άψογη διεξαγωγή των εκλογών. Ο πρόεδρος Πασινιάν τώρα θα ε, ανέλαβε στις 14 Ιανουαρίου τη θέση τα νέα του καθήκοντα ως Πρωθυπουργού και θα έχει σημαντικό έργο να ε, ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις, να προωθήσει και να ολοκληρώσει τις μεταρρυθμίσεις στην Αρμενία και σε ό,τι αφορά τα εκλογικά ζητήματα ελπίζω να ολοκληρώσει και τη μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου με βάση τη στάση του ΟΝΤΙΡ, τη δικαστική μεταρρύθμιση και την πάταξη των διακρίσεων. Θα είναι σημαντικά νομοθετήματα αυτά για το ευρύτερο δημοκρατικό κλίμα της Αρμενίας. Υπάρχουν υψηλές προσδοκίες αυτή τη στιγμή από τη νέα κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση σίγουρα θα στηρίξει τη νέα κυβέρνηση βάσει της νέας συμφωνίας που έχει τεθεί σε ισχύ, την, ε, συμφωνία, σφαιρική ε, και διευρυμένη συμφωνία εταιρική σχέση. Είχαμε την πρώτη συνδρήση της Αρμόδιας Επιτροπής 27 Νοεμβρίου που εξέτασε τον οδικό χάρτη για την εφαρμογή της νέας συμφωνίας και προσβλέπουμε στη συνέχιση των συζητήσεων για την εφαρμογή το, της συμφωνίας αυτής στο επόμενο Συμβούλιο Εταιρικής Σχέσης που θα γίνει το Μάιο ή τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πως δεν έχουμε υπόλοιπη σχόλια, οπότε μπορούμε και το σημείο αυτό, που είναι το παριθμό 7, να το κλείσουμε και να περάσουμε στο 8. Έχουμε 10 λεπτά γι' αυτό. Χωρίς λοιπόν να το καθυστερώ, η κυρία Μανέσκου ε, να μας μιλήσει για την εταιρική σχέση και τη σχετική συμφωνία με το Τουρκουμενιστάν. για τη σύναψη μιας ε, συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Τουρκμενιστάν θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω την ανακοίνωση της κυρίας Μογκερίνη πως θα ανοίξει ε, αντιπροσωπεία στο Τουρκμενιστάν η Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς, όπως, είπαμε και όπως είπα εγώ στο παρελθόν, για τον ε, φάκελο αυτό, ο δικός μας στόχος είναι η σύναψη πλήρων ε, σχέσεων με το τεκμηρισμένο στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο κράτος δικαίου, στην ενέργεια, στο κλίμα, ε, και στα πολιτικά θέματα, έτσι ώστε ο διάλογος με τα χώρα αυτή να ενισχυθεί. Θα ήθελα να εκφράσω ευχαριστίες για την πολύ αποτελεσματική προσπάθεια που κάναμε με τους ε, συναδέλφους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με τον ειδικό αποτελε... Ε, ε, τον ειδικό ε, για τις χώρες Κεντρικής Ασίας, τον κύριο Μπουριάν. Και ευχαριστώ και όλους τους συναδέλφους οι οποίοι συνεργάστηκαν μαζί μου. Υπέβαλαν πολλές ε, τροπολογίες. Την Τετάρτη που θα γίνει η συνάντηση των σκιωδών θα συζητήσουμε τις συμβαστικές προτάσεις. Το κείμενο έχει μια ισορροπία και πρόκειται να ζητήσουμε μια ξεκάθαρη διάκριση των εξουσιών ε, στη χώρα. Ζητάμε ε, και μια διαβούλευση με την Επιτροπή Βενετίας που είναι πολύ σημαντικό και ζητήσαμε να κλείσει ή το θέμα των μυστικών ε, κρατήσεων, των εξαφανίσεων και να απελευθερωθεί ε, το δικαίωμα του συνέρχεσαι να ε, επιτραπούν οι διαδηλώσεις και η ελεύθερη έκφραση των απόψεων των πολιτών. Ελπίζω πως σύντομα θα βρούμε κοινό τόπο προσπαθώντας να ορίσουμε τις ε, μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες ε, συνθήκες επί μπορούμε να συνεργαστούμε με το Τουρκμενιστάν και πιστεύω πως σε τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορούμε να αξιολογούμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί με την ε, συμμόρφωση με τα κριτήρια και να ξαναξεκινήσουμε τη διαδικασία συγκατάθεσης. Ελπίζω πως και είμαι σίγουρη πως θα συνεργαστούμε θαυμάσια και θα κλείσουμε με μια ξεκάθαρη θέση ε, με ένα πολύ χρήσιμο κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ραμόνα Μανέσκου, ήσουν σύντομοι. Ο κύριος Μπετίνη, ο κύριος Τάνοκ, όχι. Ο κύριος Σόλτς. Κύριε Μπετίνη, ξεκινάτε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το σημαντικό αυτό κείμενο που αφορά χώρα σημαντική με όλο και πιο μεγάλη στρατηγική σημασία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα έγγραφο που έχει μακρά ιστορία, το ξεκινήσαμε, το αφήσαμε, το ξαναπιάσαμε και αναφέρεται σε εγγύηση ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερίες, διάκριση εξουσιών. Κυρία Μανέσκου, η νομίζω με πολύ προσοχή και επιμέλεια παρακολούθησε την έκθεση, την επεξεργάστηκε ακούγοντας ε, και τις απόψεις των εκπροσώπων των άλλων πολιτικών ομάδων και γι' αυτό την ευχαριστώ. Σημειώνουμε βήματα πρόοδου συγκεκριμένα από φυλάκιση ορισμένων πολιτικών κρατουμένων και άρα μπορεί το Κοινοβούλιο να ε, προχωρήσει σε αποφάσεις συνενετικές ε, σημειώνω εγώ κάποιες τροπολογίες που έχω υπόψη για διευκρίνηση ή εμβάθυνση σε κάποια σημεία, αλλά πάντα βέβαια σε πνεύμα συνενετικό και συνεργατικό. Θα κατατεθούν συμβαστικά για να εξασφαλίσουμε μια γενική συνένεση στο κείμενο που θα οδηγεί στην έγκρισή του μετά. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Βετίνη. Ο κύριος Σόλτς. Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ, είναι πολύ σημαντική έκθεση. Έχει να κάνει με μια χώρα που σε σχέση με το Ουσμπεκιστάν που συζητήσαμε μόλις τώρα έχει πολύ περισσότερο περίπλοκη διαδικασία μετάλλαξης και γι' αυτό θεωρώ ε, και αυτό το απευθύνω και προς την εισηγήτρια ότι είναι πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε τι μας ενδιαφέρει στο κράτος αυτό περισσότερο. Ε, ύλε, για παράδειγμα είναι το συμφέρον μας εκεί. Πρώτε ύλε, συγκεκριμένοι πόροι που μας ενδιαφέρουν ή έχουμε και συμφέρον το ίδιο το Τουρκμενιστάν να αναπτυχθεί αυτόνομα με προοπτικές για τους πολίτες της περιοχής. Επομένως και εμείς καταθέτουμε τροπολογίες με κατεύθυνση την ε, εξισορρόπηση των πολιτικών, κοινωνικών ε, ζητημάτων, πολιτιστικών ζητημάτων κτλ. Και το ρόλο βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο να ε, συνοδεύσει το ΣΥΠΗΝ το Τουρκμενιστάν στην πορεία του αυτό ή προς τον εξυγχρονισμό. Έτσι λοιπόν ε, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη του Τουρκμενιστάν και την πρόοδό του με, την αυτό, με τον αυτοπροσδιορισμό του και βέβαια αυτό θα πρέπει να το αναζητήσουν οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι, άλλωστε όλη η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει σημασία να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια σταθερή ανάπτυξη για το Τουρκμενιστάν. Καταθέτουμε λοιπόν τι τροπολογίε μα και ελπίζουμε και εμεί, όπω είπε και η συγγήτρια, να καταλήξουμε σε ένα καλό και ισορροπημένο κείμενο που θα εκριθεί συνενετικά. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σόλτ. Άλλα σχόλια όχι. Παρακαλώ τότε τον κύριο Άιροτσεβιτς από την, από την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όντως οι αλλαγές είναι αρκετά αργές και όχι, όχι ε, τόσο φιλόδοξους όσο θα θέλαμε στον Τουρκμενιστάν. Παρ' όλα αυτά υπήρξαν κάποιες εξελίξεις που κατά τη γνώμη μου πυροδοτήθηκαν από τη συνεχή δέσμευση ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα αυτή. Τα τελευταία χρόνια και στον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με το Τουρκμενιστάν ε, έχουμε λάβει πληροφορίες από τη χώρα αυτή για πάνω από 100 υποθέσεις φυλακισμένων ή εξαφανιστέντων πολιτών και ο διαμεσολαβητής του Τουρκμενιστάν ζήτησε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη δημιουργία ικανοτήτων ε, του γραφείου του διαμεσολαβητή ε, και στην περιοχή και αυτό έγινε πέρυσι. Το Τουρκμενιστάν παίζει θετικό ρόλο και συμβάλλει στην ασφάλεια, σταθερότητα και ανάπτυξη και του Αφγανιστάν γιατί οι δύο χώρες έχουν ε, κοινά σύνορα μήκους 750 χιλιόμετρων και είναι προ όφελό μα να στηρίξουμε τις προσπάθειες ε, του Τουρκμενιστάν στο Αφγανιστάν. Γιατί οποιαδήποτε αποσταθεροποίηση τη κατάσταση στα σύνορα μεταξύ των δύο χωρών θα χρησιμοποιηθεί από τρίτε χώρε. Υπήρξαν κάποια κάποιε θετικέ ενδείξει σταδιακή μετάβαση του Τουρκμενιστάν στην οικονομία τη αγορά. Κάτι που θα δημιουργήσει περισσότερε ευκαιρίε για περισσότερε ε, συναλλαγέ με τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει ε, για παράδειγμα, ε, σχέδια για ιδιωτικοποίηση του ξενοδοχειακού κλάδου και του ελευτικού κλάδου στο Τουρκμενιστάν. Βέβαια, θα υπάρξουν πολλές ευκαιρίες ε, σχέσεων ε, με τους διάφορους μηχανισμούς της κυρωμένης συμφωνίας θερικής σχέσης και συνεργασίας, κάτι που θα φέρει αρκετούς καρπούς. Στην περίπτωση του Σμπεκιστάν διαπιστώσαμε ότι πολλές θετικές αλλαγές ε, κατέσαν δυνατές και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για ενισχυμένη, διευρυμένη συνεργασία εν αυτό το χρόνο. Και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα συνεχίσει να τροφοδοτεί με πληροφορίε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη συνεργασία και την πρόοδο που σημειώνουμε στη σχέση μα με το Τουρκμενιστάν και ιδιαίτερα στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και μπορώ να σας επιβεβαιώσω ότι στόχος μας είναι ε, το άνοιγμα ενός γραφείου στο Τουρκμενιστάν μιας ε, κανονικής αντιπροσωπείας στη διάρκεια του 2019. Αφού δεν υπάρχουν άλλα σχόλια λοιπόν, να σας ενημερώσω και πάλι. 4 Φεβρουαρίου ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ και ελπίζουμε να ψηφίσουμε σε κάποιο ολομέλεια του Μαρτίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ραμόνα για όσα, τα μας, για όσα μας είπες και μπορούμε τώρα να περάσουμε στα σημεία 9, 10, 11 και 12 Ελπίζω οι προσκεκλημένοι μας να είναι ήδη εδώ και θα συνεχίσουμε σε ένα λεπτό. Anyone So, colleagues, we come to items number... Αγαπητοί συνάδελφοι, περνούμε στα σημεία 9, 10, 11 και 12 που στο σύνολό τους αφορούν το Αφγανιστάν. Δεν σας διαβάζω τους τίτλους όπως προβλέπονται. Βλέπετε ότι υπάρχει εμβάθυνση των σχέσεων, αλληλεγγύη, μακροχρόνιες σχέσεις με το Αφγανιστάν, συμφώνια εταιρική σχέση του Φεβρουαρίου του 2018, που περιμένει κύρωση από το Κοινοβούλιο, διάσκεψη στη Γενέβη τέλη Νοεμβρίου του 2018 για να επιβεβαιωθούν αμοιβαίες δεσμεύσει τη διεθνού κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κοινοβούλιο υποστηρίζουν αυτέ τι μεταρρυθμίσει και τι προσπάθειε για την αλληλεγγύη, την διαμεσολάβηση και την οικονομική υποστήριξη. Προχωρούμε σε ανταλλαγή θέσεων και απόψεων για την κατάσταση στην χώρα, ενωπιώντας όλα τα θέματα αυτά της της διάταξης. Πρώτη είναι η κυρία Πάολα Παμπαλώνη, αν δεν κάνω λάθος στην προφορά του ονόματό τη, η οποία αντικαθιστά τον ειδικό απεσταλμένο για το Αφγανιστάν, κύριο Κόμπια, ο οποίο, όπω είπα, είχε κόλλημα λόγω επίγουσων υποχρεώσεων και δεν μπόρεσε να έρθει. Θα ακούσουμε λοιπόν την κυρία Παμπαλώνη, στη συνέχεια τον κύριο Άουστρεβιτσιους για την επίσκεψη της αντιπροσωπείας μας στην Καμπούλ πριν τα Χριστούγεννα και εν τέλει σχέδιο νομοδότησης με 24 συμβιβαστικές τροπολογίες για την εταιρική σχέση και ανάπτυξη μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισλαμική Δημοκρατία του Αφγανιστάν. Η κυρία Παμπαλώνη, λοιπόν, παρακαλώ να λάβει το λόγο. Και καλώ ήρθατε στην σπουδαιότερη Επιτροπή του Κοινοβουλίου, την ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την πρόσκληση αυτή στην ε, Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας για την θετική αξιολόγηση στο σχέδιο έκθεσης για την συγκατάθεση στην ε, συμφωνία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν. Ήμουν η διαπραγματεύτρια στην ε, συμφωνία αυτή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και χαίρομαι που συνέβη αυτό και που παραβρέθηκα σε αυτή την συγκατάθεση από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολύ καιρό διαπραγματευόμασταν. Την εντολή από το Συμβούλιο τη λάβαμε τον Νοέμβριο του 2011. Πολλά χρόνια διαπραγματεύσεων με κάποιες διακοπές και στις τελευταίες εκλογές και μετά ξαναξεκινήσαμε με τη νέα κυβέρνηση και επιτέλους υπεγράφει στις 18 Φεβρουαρίου του 17. Ε, είπατε εκπρόσωπος κυρία Μεγκυρίνη υπέγραψε τη συμφωνία αυτή. Ήθελα να σας κάνω ένα briefing για το πού βρισκόμαστε σήμερα και να σας πω ποια είναι η σημασία της συμφωνίας αυτής στις διμερείς σχέσεις που έχουμε μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφγανιστάν. Καταρχήν, είναι το μοναδικό νομικό ε, πλήρες πλαίσιο το οποίο ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ Αφγανιστάν και Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε ήδη θέσει σε προσωρινή εφαρμογή τη συμφωνία αυτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια σειρά συναντήσεων στα πλαίσια της ε, συμφωνίας αυτής. Η Μικτή Επιτροπή στα πλαίσια της προσωρινής εφαρμογής συνεδρίασε για πρώτη φορά πέρυσι και είχαμε και την πρώτη συνεδρία της Ομάδας Εργασίας για την Χρηστή Διαχείριση των ανθρώπινων Δικαιώματα και τη Μετανάστευση αυτές οι δύο συναντήσεις ήταν πάρα πολύ σημαντικές γιατί έχουμε μια σειρά θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τις μεταξύ μας σχέσεις και τα οποία συζητήσαμε με ανοιχτό και με επικοδομητικό τρόπο. Δηλαδή, Μιλήσαμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ισότητα των φύλων, για την αναπτυξιακή βοήθεια, το εμπόριο, τις επενδύσεις, την περιφερειακή συνεργασία, τη μετανάστευση και κάναμε και μία απογραφή της τρέχουσας κατάστασης, πρόοδου που έχει σημειωθεί και πιο συγκεκριμένα ποιες είναι οι ε, προκλήσεις που είναι σε εκκρεμότητα έτσι ώστε να υποβάλουμε κάποιες συστάσεις. Εμείς παρακολουθούμε συνέχεια την κατάσταση και μετά τις δύο αυτές συναντήσεις. Είμαστε επίσης στη διαδικασία προετοιμασίας του επόμενου γύρου συναντήσεων και στις συζητήσεις μας που θα κάνουμε με τις Αυγανικές αρχές το 19 θα σας ενημερώνουμε συνέχεια για κάθε εξέλιξη. Καλωσορίζουμε τώρα την πλήρη επικύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας από όλα τα κράτη-μέλη. 15 το έχουν ήδη πράξει και περιμένουμε όπως σας είπα και τους ε, υπόλοιπους όπως επίσης και στη συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλα τα θέματα που καλύπτει η συμφωνία αυτή έτσι ώστε να μπορούν ε, να τεθούν και αυτά υπό τούτο το νομικό πλαίσιο. Στις διμερείς ε, επαφές που έχουμε, έχουμε δύο βασικά στρατηγικά έγγραφα. Ένα είναι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για το Αφγανιστάν, που εγκρίθηκε το 17 από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και τα πιο πρόσφατα συμπεράσματα του Συμβουλίου από τον Νοέμβριο του 2018. Οι σχέσεις μας με το Αφγανιστάν θα μπορούσαν ε, να περιγραφούν ως εξής. Το πιο σημαντικό πολιτικό θέμα το οποίο έχουμε στα πλαίσια του διαλόγου είναι η πρόθεση της ειρήνης, της σταθερότητας και της περιφερειακής ασφάλειας. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι της στρατηγικής μας. Δεύτερον, η ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πιο συγκεκριμένα η πριόθεση ε, και η χειραφέτηση των γυναικών. Τρίτον, στήριξη την οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη και τέλος, αλλά όχι ίσονος σημασίας, οι προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση ε, και τις εξαναγκαστικούς ε, ε, εκτοπισμούς που είναι ένα θέμα ακόμα στο Αφγανιστάν. Ενισχύουμε αυτή τη στιγμή τη διμερή μας σχέση με την κυβέρνηση και ενισχύεται και η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Συστάμε πολλά θέματα μεγάλη γκάμα. Δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, μεταρρυθμίσεις, ειρήνευση και ποιο είναι ο συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει στη διαδικασία ειρήνευση. Στα πλαίσια του διαλόγου μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τόνισε τη σημασία που έχει το να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και κυρίω η μάχη για την πάταξη τη διαφθορά, υπέρ του κράτου δικαίου, πολύ σημαντικά θέματα ε, που θα συνεχίσουν τα όσα έχουμε κάνει ε, με τις αποστολές μας εκεί, όπως επίσης και η μεταρρύθμιση ε, της δικαιοσύνης, για να δούμε και το θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών. Συμπέρασμα. Σε πολλούς χώρους έχουμε δει μεγάλη πρόοδο με νέα νομοθεσία που αυτή τη στιγμή συντάσσεται, η οποία είναι πολύ ικανοποιητική. Όμως, η μεγάλη πρόκληση μπροστά μας είναι πώς η νομοθεσία αυτή θα εφαρμοστεί και αυτό βέβαια σε σχέση με το τι λένε οι διεθνείς κανόνες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες έτσι ώστε να εκπαιδεύσουμε την διοίκηση και την κυβέρνηση για το πώς η νομοθεσία αυτή θα εφαρμοστεί και να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση του πληθυσμού για την νομοθεσία η οποία προσφέρει σημαντικά δικαιώματα στις πιο ευάλωτες ομάδες του χώρα. Το θέμα στο οποίο είμαστε ιδιαίτερα παρόντες στο Αφγανιστάν αυτή τη στιγμή είναι, και θα ξεκινήσω με τη μάχη για την πάταξη της διαφθοράς, εμείς Κάθε χρόνο οργανώνουμε μια μεγάλη συνδιάσκεψη για κατά της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο. Το κάναμε πέρσι τον Απρίλιο και θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να οργανώσουμε κάτι αντίστοιχο φέτος έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί η κυβέρνηση, η δίκτυα και ο πληθυσμό για το τι δράσεις χρειάζονται να αναλυφθούν για τη μάχη κατά της διαφθοράς. Δεύτερον, προσπαθούμε να βοηθήσουμε την κυβέρνηση και τις ε, ανεξάρτητες αρχές για να προετοιμάσουν τις εκλογές. Έγιναν κοινοβουλευτικές εκλογές ε, τον Οκτώβριο με καλά θέματα και πρέπει να σας πω ότι οι νέοι και οι γυναίκες συμμετείχαν ε, στις εκλογές αυτές, αλλά είχαμε και λήψεις και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να ξεπεράσει αυτές τις δυσκολίες εν ώψη της προετοιμασίας της πιο σημαντικής εκλογής που είναι η προεδρική που θα γίνει 20 Ιουλίου του 19. Έχουμε μια σειρά project τα οποία εφαρμόστηκαν μαζί με την κυβέρνηση και την ε, αποστολή των Ηνωμένων Αθνών για να στηρίξουμε την εκλογική διαδικασία έτσι ώστε να ενισχυθεί η ε, νομιμοποίηση και της κυβέρνησης και της Προεδρίας μετά τις εκλογές. 15 εκατομμύρια ευρώ έχουμε διαθέσει στην αποστολή των Ηνωμένων Αθνών, στην Ουνάμα και έχουμε και βοήθεια προς την κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να ευαισθητοποιηθεί ο πληθυσμός να γνωρίζει πως γίνεται αυτή η εκλογική διαδικασία και εδώ η χρηματοδότηση είναι ε, αυτό που σας είπα, είναι 3,5 εκατομμύρια για την ειρηνευτική διαδικασία. Ε, μεταρρυθμίσεις στην αστυνομία διάλογος εκεί με την κυβέρνηση. Έχουμε ένα project το οποίο αποτελείται από 10 συμβούλους στο Υπουργείο Εσωτερικών και στην αφγανική αστυνομία η οποία προσπαθεί, ε, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν να βοηθήσουν την αστυνομία ε, να δημιουργήσει και μία ε, πολιτοφυλακή και επίσης πιο σημαντικό να εκπαιδεύσει και γυναίκες αστυνόμους. Μετανάστευση. Εδώ συνεργαζόμαστε πολύ με την τη Γενική Διεύθυνση ΤΕΒΚΟ και τους συναδέλφους από την Κομισιόν. Έχει ξεκινήσει ένας μεγάλος διάλογος με το Αφγανιστάν για τη μετανάστευση, με κάποια έγγραφα τα οποία αποτέλεσαν την εκκίνηση του διαλόγου για την εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής παρανόμων μεταναστών που βρίσκονται στην Ευρώπη και δεν, περιμένουμε, δεν παραμένουμε εκεί. Χάρη στη Συμφωνία Συνεργασίας έχει ξεκινήσει και διάλογος για τη μετανάστευση η οποία ε, γίνεται σε περιφερειακό πλαίσιο, δηλαδή προκλήσεις που αντιμετωπίζει το Αφγανιστάν με την επιστροφή προσφύγων ε, από το Αφγανιστάν που έχουν καταφύγει στο Ιράν και στο Πακιστάν και εκεί έχουμε προσφέρει πολλά χρήματα για την επανένταξη αυτών των ε, ε, προσφύγων που επιστρέφουν. Επίσης παρακολουθούμε πολύ στενά τις εξελίξεις στο Πακιστάν και οι τελευταίες προφορίες που έχουμε μετά τις δηλώσεις του κυρίου Καν, που είναι ο Πρωθυπουργό του Πακιστάν, είναι η δυνατότητα του να δοθεί πακιστανική υπηκότητα στους Αυγανούς που έχουν γεννηθεί στο Πακιστάν. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη. Εφόσον βέβαια γίνει πράξη. Τέλος για το θέμα της ειρηνευτικής διαδικασίας. Ε, καταρχήν, ο κύριος Κοπίες θέλει πάρα πολύ να έρθει κοντά σας σήμερα και να σας ενημερώσει για το τι γίνεται με την ειρηνευτική διαδικασία. Είναι έτοιμος να έρθει σε μια επόμενη συνεδρίαση της ΑΦΕΤ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Καμπούλ για να συζητήσει με τον πρόεδρο και τους εμπλεκόμενους τη συγκεκριμένη εφαρμογή της προσφοράς που έκανε η κυρία Μογκερίνη στη Γενέβη στην Υπουργική Διάσκεψη πέρυσι, όπου είπε υπάρχουν πέντε σημεία στα οποία μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει ε, να στηρίξει την ειρηνευτική διαδικασία. Και τι είπε, είπε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ανοίξει την ειρηνευτική διαδικασία, μπορούμε να στηρίξουμε μπορούμε να βοηθήσουμε με τις μεταρρυθμίσεις και κυρίως στον ε, χώρο των δυνάμεων ασφαλείας. Να στηρίξουμε επίσης τρίτον την επανένταξη των πρώην πολεμιστών και των οικογενειών τους, έτσι ώστε να επανενταχθούν στην κοινωνία, στην εργατική, στο εργατικό δυναμικό. Τέταρτον, να είναι εγγυητής η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια επόμενη συμφωνία ειρήνευσης στο Αφγανιστάν. Και τέλος, πέμπτο σημείο, προσέφερε να ενισχύσει την προώθηση της περιφερειακής, ε, του περιφερειακού εμπορίου και των περιφερειακών υποδομών. Πολύ σημαντικά αυτά τα οποία ε, προσέφερε η Πατή Εκπρόσωπος και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να γίνουν πράξη. Αυτή τη στιγμή ο ειδικό απεσταλμένος είναι στην Καπούλη για να συζητήσει όλα τα θέματα αυτά. Αυτά. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστούμε κυρία Παμπαλόνη, για την ενημέρωση. Θα ήθελα πρώτα να ρωτήσω τον Τσάρλ Στάνοκ. Θέλεις να πεις κάτι εκ μέρους της κυρίας Φωτίκα που απουσιάζει, ναι. Μου έχει δώσει τη δήλωσή της να της τη διαβάσω. Για τους συναδέλφους που δεν ήταν πριν ε, για να ακούσουν ε, απουσιάζει λόγω ασθένειας η κυρία Φωτίγκα, η συγγετρία. Δεδομένου, λοιπόν τη συμφωνία συνεργασία, ε, μάλλον τη εταιρική σχέση για τη συνεργασία και την ε, ανάπτυξη του Αφγανιστάν, είναι το πρώτο νομικά δεσμευτικό πλαίσιο για τι σχέσει μα με τη χώρα αυτή. Η έκθεση κάνει ένα απολογισμό τη κατάσταση ε, και ε, ζητά βιώσιμες πολιτικές για να εξασφαλιστεί το, η αξιοποίηση του δυναμικού των σχέσεων από την αναπτυξιακή βοήθεια, συνεργασία για την αντιτρομοκρατία και την ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικές όπως γεωργία, περιβάλλον και η δημόσια υγεία. Επίσης θέλουμε να στηρίξουμε την κοινωνία των πολιτών αξιοποιώντας τα θεωρητικά σημάδια που έχει δείξει ε, ε, το Αφγανιστάν σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση ικανοτήτων και την κατάρτιση των δυνάμεων ασφαλεία. Ε, από την απόσυρση του διεθνών δυνάμεων το 2014 ξεκίνησε μια μεταβατική περίοδος και καλό θα ήταν να συνεργαστούμε με το Αφγανιστάν και τους ομοιδιάτες εταίρους μας για να αντιμετωπίσουμε τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Επίσης, να μην ξεχνούμε και την ευθύνη των γειτονικών χωρών και των περιφερειακών δυνάμεων για να δημιουργηθεί ένα ασφαλέ και σταθερό Αφγανιστάν. Μόνο έτσι θα εξασφαλιστεί ένα ευημερό μέλλον και για το Αφγανιστάν αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά και σα ευχαριστώ εκ μέρου τη συγκεκριτής κυρία Φωτίγκα. Ευχαριστώ τώρα ο Πέτρα Αυστρεβίτσιος θα μα κάνει την ενημέρωση από την πρόσφατη αποστολή μα στην Καμπούλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Παμπαλώνη, ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση που μας κάνατε για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και τις σχέσεις μας. Όπως είπε και ο πρόεδρος στην αρχή, πριν τα Χριστούγεννα μετέβημε στο Αφγανιστάν και δεν πήγαμε αναζητώντας τον Άγιο Βασίλη. Ξέρουμε που ζει ο Άγιος Βασίλης. Ήταν μια ειδική αποστολή και ο Αντρέα Έλισον και ο Φρανκ Έγγελ με συνόδευσαν σε αυτή την ειδική αποστολή που πραγματοποιήσαμε στο Αφγανιστάν και λόγω ρυθμίσεων ασφαλείας που είναι πολύ αυστηρές για το Αφγανιστάν είχαμε απλώ την ευκαιρία να παραμείνουμε στην Καμπούλ ε, και να επισκεφτούμε μόνο κάποια ε, κυβερνητικά κτίρια και τους ειδικού ε, χώρους για τους οποίους είχαμε πάρει άδεια. Υπάρχει μια αίσθηση κόπωσης ε, στο Αφγανιστάν. Αυτό είναι ένα γενικό συμπέρασμα. Και ο λαός απεγνωσμένα ζητά ειρηνευτικές λύσεις, γιατί δεν υπάρχει στρατιωτική λύση για το Αφγανιστάν και αυτό είναι σαφές. Αυτό το έχουν πια συνειδητοποιήσει οι πάντες. Αλλά θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το Αφγανιστάν στη μοίρα του, όπω τώρα. Η θα δούμε έξαρση νέων τρομοκρατικών δυνάμεων και ανάπτυξη νέων τρομοκρατικών ομάδων που θα επεκταθούν στο Αφγανιστάν δημιουργώντας μια κατάσταση που δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή ούτε καν να τη συλλάβουμε. Συναντήσαμε πολλούς υψηλούς αξιωματούχους, τον πρόεδρο Γκανή, τον Αμπτούλα Αμπτουλά, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον πρώην πρόεδρο Καρζάη, πολλούς ε, υψηλά ιστάμενους και πολιτικούς ηθήνοντες. Ενημερωθήκαμε λοιπόν εκτενώς για την κατάσταση στο Αφγανιστάν και θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια σημεία από τις συζητήσεις μας. Την ημέρα της αύξησης μας ε, ξεκίνησαν σχεδόν την ίδια μέρα οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ταλιμπάν και των εκπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και η επίσημη αντιπροσωπεία του Αφγανιστάν δεν έλαβε άδεια να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία, δυστυχώς. Οπότε υπήρχε υπάρξει αίσθηση ότι δεν ήταν ουσιαστικέ και γνήσιε οι διαπραγματεύσει, ε, παρόλο που όλοι δήλωσαν ότι αναζητούν μια ειρηνευτική λύση. Ακούσαμε όμω από πολλού πολιτικού και από καλά κατατοπισμένου για την κατάσταση ότι δεν θα πρέπει ε, μια απλή ειρήνη να έχουμε στο Αφγανιστάν, αλλά ειρήνη χωρίς αποκλεισμούς που θα λαμβάνει υπόψη όλα τα μέχρι τώρα επιτεύγματα της διαδικασίας. Δηλαδή θα εξασφαλίσει την πλήρη συμμετοχή και των γυναικών στο δημόσιο βίο, στην παιδεία επίσης ε, που θα πρέπει να συνεχιστεί και φυσικά να αξιοποιηθούν όλα τα μέχρι τώρα επιτεύγματα για τη δημιουργία των κρατικών θεσμών. Αλλά αυτά θα πρέπει να διασφαλιστούν. Όχι η ειρήνη πάση θυσία λοιπόν, αλλά συγκεκριμένε προδιαγραφέ. Παρ' όλα αυτά, και για όλου αυτού του λόγου, μάλλον είναι κάπω αόριστη η κατάσταση και κάπω αμυδρέ οι προοπτικέ της Ειρήνη. Συναντηθήκαμε και με τον πρόεδρο των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν και πραγματικά <laughs> έχουμε πολλού διπλωμάτε Αμερικανού στην Καμπούλ ε, και τους ζηλεύω γιατί είναι πολύ καλά εξοπλισμένοι και έχουν εγκατασταθεί θαυμάσια. Μακάρι και η δική μας αντιπροσωπεία, η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει κάτι αντίστοιχο αμυδρά αντίστοιχο με αυτά που απολαμβάνουν οι Αμερικανοί διπλωμάτες στην Καμπούλ. Και νομίζω ότι θα πρέπει να μετακομίσουμε ε, γιατί λόγω των ρυθμίσεων ασφαλείας είναι πολύ χρονοβόρη μετα... μετακίνησή μας στην Καμπούλ για τη συναντήση με υψηλά ισταμένους. Δεν είναι εύκολη, εύκολη πρόσβαση, οι, οι δρόμοι είναι γεμάτη κόσμο, πολλές φορές δημιουργείται κυκλοφοριακή συμφόρηση, είναι δύσκολο να περάσει κανείς και δεν είναι ασφαλές ε, για οποιοδήποτε αξιωματούχο να επισκέπτεται την Καμπούλ και το Αφγανιστάν και να κινείται ελεύθερα. Οπότε θα πρέπει να ζητήσουμε καλύτερη ε, τοποθέτηση, καλύτερο εξοπλισμό των δικών μας διπλωματών στην Καμπούλ, αντίστοιχα με αυτό που λαμβάνουν οι Αμερικανοί διπλωμάτες. Και Κάποια άλλα πολύ σημαντικά θέματα αφορούν την εκλογική διαδικασία, για παράδειγμα. Δεν έχουμε λάβει ακόμη τα τελικά, τα οριστικά αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών που έγιναν στο Αφγανιστάν. Είναι πολύ χρονοβόρα, πολύ αργή διαδικασία. Δυστυχώ ακούστηκαν πολλέ επικρίσει ε, για τη διαδικασία αυτή λόγω διαφάνεια κλπ. κλπ. είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ε, παγκόσμιος εταίρος και θα πρέπει να λάβει ιδιαίτερη θέση στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και προσβλέπω στην αναβάθμιση του ρόλου μας και της θέσης μας εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Δύο σκιώδεις ηγητές, και Βαλέρο, έχουν ζητήσει το λόγο. Α, όχι. Μ, λάθος πληροφορία. Κυρία Βαλέρο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας, θα μιλήσω σου ειδικά. Σας άκουσα με πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε χρόνο πιστεύω ακόμα. Έχουμε πολλή δουλειά μάλλον για να εξασφαλίσουμε βιώσιμη λύση στο Αφγανιστάν. Πρέπει να ξαναχτιστεί η χώρα, να εξασφαλιστεί η οικονομική ανεξαρτησία, αυτονομία, ο σεβασμός των μειονοτήτων όποιες και είναι αυτές, δεν είναι δεδομένο σήμερα και πρέπει να συνεχίσει σε αυτή την πορεία. Ιδιαίτερα σε σχέση με την κοινωνία των πολιτών. Λυπηρό στην πολιτική μας σε σχέση με το Αφγανιστάν είναι το ότι εδώ στην Ευρώπη συζητούμε κυρίως τις ε, συμφωνίες επανεισδοχής ή ε, επανόδους του Αφγανιστάν που συστούμε εδώ και χρόνια, που όμως ξέρουμε ότι η κατάσταση στη χώρα είναι τόσο δύσκολη και περίπλοκη που πράγματι αντιμετωπίσουν πολλά προβλήματα οι νεαροί Αφγανοί που μπορεί να στέλνουν πίσω στην πατρίδα τους σε μια χώρα που δεν έχει τα μέσα να τους υποδεχθεί. Καλά και αν τους στέλναμε μόνο εμείς οι Ευρωπαίοι μπορεί να ήταν διαφορετικό το πρόβλημα αλλά είναι εκατομμύρια οι Αφγανοί που έχουν βρει καταφύγιο σε γειτονικέ χώρες και κινδυνεύουν και αυτοί να ε, αναγκαστούν να επιστρέψουν στη χώρα τους, ενώ η χώρα, το Αφγανιστάν, δεν τα καταφέρνει, δεν μπορεί να τους ε, υποδεχθεί. Πρέπει να βρούμε μια λύση λοιπόν στην Ευρώπη και να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις ε, επανειστοχές ή στις απελάσεις. Πρέπει να δούμε τι συμβαίνει στην ε, πραγματικότητα. Οι νέοι όταν έρχονται εδώ στις χώρες μας πρέπει να έχουν την ευκαιρία για κατάρτιση, για εκπαίδευση και να μπορούν επιστρέφοντας στη χώρα τους καταρχάς να το θέλουν και δεύτερον να είναι σε θέση να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση της χώρας. Έχουμε λοιπόν μια μελέτη σε ένα φυλάδιο του Save the Children, σωστά τα παιδιά που δείχνει τι παθαίνουν τα παιδιά αυτά, τι περνούν. Πρέπει να το διαβάσετε για να καταλάβουμε τι συνέπειες έχει το να στέλνουμε πίσω είτε ενήλικες είτε και παιδιά στη χώρα αυτή. Αντιμετωπίζουν τη βία, αντιμετωπίζουν την ε, ε, επιστράτευση από διάφορες ε, παραστρατικές οργανώσεις. Ε, πάση περιπτώσει θα θέλω να ευχαριστώ την κυρία Φωτσίγκα που έκανε δεκτές τις τροπολογίες μας και θα ήθελα να πω και εγώ ότι ήταν εξαιρετική συνεργασία. Ευχαριστώ κυρία Βαλέρο, κύριο Λαλόντ. Κυρία Λαλόντ, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Καταρχάς ευχαριστώ τον συναδελφό Μοσκοβίτσους για την έκθεσή του και για την επίσκεψη στην Καμπούλ. Δεν είναι καθόλου απλά τα πράγματα εκεί. Εγώ γνωρίζω τη χώρα καλά γιατί 15 χρόνια πηγαίνω τακτικά. Και όχι μόνο στην Καμπούλ, αλλά και στο βορρά. Και πρέπει να πω ότι αισθάνομαι επιφυλακτικότητα 18 χρόνια τώρα που έχει απο... απελευθερωθεί από τους Ταλιμπάν το, το Αφγανιστάν και ύστερα από μια πολύ σημαντική περίοδο ελπίδων ε, μεταξύ 2003-2008 λίγο πολύ όπου μπορούμε να πούμε άνθησε το Αφγανιστάν ε, οι γενικές εκλογές είχαν μάλιστα οδηγήσει 23 23% ε, γυναίκες να αναλάβουν ε, καθήκοντα στα έδρανα του Αφγανικού Κοινοβουλίου. Οι φίλοι και οι φίλες που έχω στο Αφγανιστάν, ε, έμπλεοι, εξυγχρονισμού, τα πράγματα φαίνονται να πηγαίνουν καλύτερα, τα παιδιά πήγαιναν στο σχολείο κτλ. Και από τη στιγμή που έχει αρχίσει μια προσπάθεια για διαπραγμάτευση με του Ταλιμπάν, βλέπω και περισσότερες επιθέσεις να γίνονται και να επιδεινώνεται η κατάσταση στη χώρα. Τώρα βλέπω να υπάρχει μια προσπάθεια για επιδίωξη συνομιλιών. Δεν το υποστηρίζω επουδενή. Δεν πιστεύω καθόλου ότι μπορεί να προστατέψουν όπως μπορεί να ισχυρίζονται οι Ταλιμπάν τα δικαιώματα των γυναικών, γιατί ξέρω ότι σε δύο-τρία χρόνια θα αντιστραφεί η κατάσταση ριζικά. Και θεωρώ ότι αυτή η επαφή με τους Ταλιμπάν ε, θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. για τις προεδρικές εκλογές έχουμε πάνω από 10 υποψηφίους, τον ε, τωρινό πρόεδρο Ασραπναβή, τον Απτουλά Απτουλά, που έχει την υποστήριξη του αντιπρόεδρου Ντασραμγκάνη, του Ντασραμγκάνη που είναι ο Ντόξτομ. Δεν θα σας πω το όνομα των όλων ε, των βουλευτών, αλλά υπάρχει ο Μασούτ, και άλλοι, άλλος επικεφαλής ε, της Μυστικής Υπηρεσίας, ο Φατσνά. Σοβαρή υποψήφη, πολύ καλά. Και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει ό,τι μπορεί για να δώσει ένα πλαίσιο για αυτή την ανταμέτρηση. Αυτά ήθελα εγώ να μοιραστώ μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν είστε κανείς άλλο στο λόγο. Ο κύριος Ιόντιτσε από τη Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξιακής Συνεργασίας και μετά εσείς κυρία Παμπαλόνια. Κυρία, παρακαλώ. Εδώ είμαι. Και θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα είπε η συνάδελφος Πάολα. Διαβάζουμε με μεγάλο ενδιαφέρον την έκθεση του Κοινοβουλίου και συμμεριζόμαστε τις ε, παρατηρήσεις του. Η Επιτροπή με τα της ε, ταμεία έχει αναλάβει ε, η δράση, έχει αναπτύξει δράση διάφορους τομείς και αξιολογήσαμε τις πρόοδους που προκύπτουν σε συνεργασία με την κυβέρνηση και τη στράτευση της, την προσήλωση της μεταρρυθμίσης. Μία από τις φράσεις που έχει χρησιμοποιήσει ο πρόεδρος του Αφγανιστάν ήταν ότι οι Ευρωπαίοι κρατάνε το χρονόμετρο, το Αφγανιστάν κρατάει το χρόνο. Δηλαδή ότι χρειάζεται χρόνος για να φτάσουμε στα αποτελέσματα. Επίσης, ε, δραστηριότητα αναπτύχθηκε και στο πεδίο της μετανάστευσης, στην Σύνοδο της Γενέβης, υποδομές, που υπογραμμίζουν τη σημασία των περιφερειακών παραγόντων στον διάλογο αυτό για την ειρήνη, για το Αφγανιστάν και υποστηρίξαμε την χορήγηση 572 εκατομμυρίων ευρώ για το Αφγανιστάν στη Γενέβη. Επίσης, ειρήνη, ε, ανοικοδόμηση των κρατικών δομών, μεταρρυθμίσεις για την πάταξη της διαφθοράς, Το 2016 ξεκινήσαμε με βάση τον προϋπολογισμό μία προσέγγιση, δηλαδή με, τις, με στοχευμένες συμβάσεις, αλλά με διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν και με το περιβάλλον και με την αγορά εργασίας, με τη δημοκρατία και τα λοιπά εμπειρίες που οδηγούν σε μια νέα συμφωνία για 300 εκατομμύρια για την ανεκοδόμηση και την ε, οικοδόμης εμπιστοσύνη. Και ε, θα ήθελα να τονίσω πέραν των όσων είπε η συνάδελφο ότι τα αναπτυξιακά αυτά μία ιδιαίτερα απευθύνονται σε νέου που επανέρχονται από γειτονικέ χώρε, Ιράν, Πακιστάν και άλλε, και όχι μόνο από την Ευρώπη, αλλά απευθύνεται και σε εσωτερικώ εκτοπιστέντε. Προσβλέπουμε στην περαιτέρω συνεργασία, στο διάλογο για την ειρήνη, όπως άλλωστε εξήγησε και η Υπηρεσία Εξωτερικής δράση Νωρίτερα, ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Παμπαλώνη για την ολοκληρώση της Θα είμαι πάρα πολύ ε, σύντομη. Ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχετε θίξει που σχετίζεται και με το κόστος της ειρήνευσης και με την στήριξη που προσφέρουμε εμείς. Εμείς θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε και προσπαθούμε να διαβεβαιώσουμε και τις γυναίκες του Αφγανιστάν πως η διαδικασία ειρήνευσης ε, δεν πρόκειται να επιδιωχθεί ε, όποια και να είναι η τιμή αυτή. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διατηρήσουμε όλες τις προόδους και τις, ε, τα κέρδη που έχουμε πετύχει τα τελευταία 17 χρόνια και επιβεβαιώνω πως οι γυναίκες στο Αφγανιστάν εκφράζουν το φόβο πως ο διάλογος με τους Ταλιμπάν και η διαδικασία ειρήνευσης μπορεί ως αποτέλεσμα να μειώσει ή και να ακυρώσει τα δικαιώματα τα οποία έχουν πετύχει με τόσες δυσκολίες ε, στα χρόνια αυτά οι γυναίκες. Ένα λοιπόν από τα ισχυρά μηνύματα τα οποία κατατέθηκε στην ε, διάσκεψη της Γενέβης είναι πώς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τη διαδικασία ειρήνευσης, πού θα προκύψει το διάλογο αυτό, αλλά υπό την προϋπόθεση πως τα θεμελιώδη ε, δικαιώματα και κυρίως αυτά των γυναικών τα οποία αποκτήθηκαν μέχρι σήμερα θα διατηρηθούν στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι σημαντικό και είναι σημαντικό να ακουστεί η φωνή μας και αυτό να γίνει και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το βλέπω και σε πολλά από τα δικά σας ψηφίσματα είναι λοιπόν ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει με τον τρόπο αυτό στην ειρηνευτική διαδικασία. Επίσης, ένα σημαντικό βήμα ακόμα είναι η επόμενη συνάντηση στη διαδικασία της Καμπούλ, 28 Φεβρουαρίου. Εκεί θα συνεργαστούμε με την κυβέρνηση και όσους προσπαθούν να διευκολύνουν την ειρήνευση για να είμαστε κι εμείς παρόντες, για να έχουμε κι εμείς μια φωνή στον επόμενο γύρο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Παμπαλώνη. Δεν έχουμε λοιπόν άλλα σχόλια από ό,τι βλέπω. Θέλω να σας ενημερώσω πως η Επιτροπή θα ψηφίσει αύριο το πρωί και στην Ολομέλεια θα περάσουμε την πρώτη Ολομέλεια του Μαρτίου. Σας εύχομαι καλό βράδυ εσάς κυρία μου, εμείς έχουμε και άλλα ακόμα θέματα στην ημερήσια διάταξη. Είμαστε στο 13, ανταλλαγή απόψεων για μια πρωτοβουλία ε, για το τι θα συμβεί στην περιοχή ΜΕΒΑ για την ε, περίοδο μετά την Αραβική Άνοιξη, οπότε επειδή έχουμε καθυστερήσει, κύριε Μπενιφέη, στο εισηγητή μας για δεύτερη φορά σας δίνω το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Οχτώ χρόνια μετά τις ε, λεγόμενες αραβικές ανοίξεις ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στις εξελίξεις και τη δράση βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αξιολογήσουμε τα θετικά στοιχεία και να ενθαρρύνουμε ε, τις αλλαγές ε, σε σχέση με τα αρνητικά. Ιδιαίτερα στεκόμαστε στα άτομα νέοι άντρες και γυναίκες σε εκατομμύρια που βγήκαν στους δρόμους το 2011 σε μεγάλο μέρος των κρατών αυτών ζητώντας καλύτερες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, αξιοπρέπεια, συμμετοχή στο δημόσιο βίο και στην κοινωνία τους. Όπως ξέρουμε, οι επιλογές των διαφορών κρατών ύστερα από, και οι πορείες των κρατών αυτών ύστερα από τα γεγονότα ήταν διαφορετικές ανάλογα το κράτος από την ε, πορεία προς την εκδημοκρατία ε, μέχρι τη δημοκρατία, αλλά ακόμα και τον εμφύλιο πόλεμο, του οποίου τις συνέπειες ακόμα ζούμε. Ε, βλέπουμε επίσης ότι υπήρξε μια προσπάθεια εκδημοκρατισμού, αλλά παραμένουν προβλήματα, όχι μόνο κοινωνικό-οικονομικά. Προβλήματα που απαιτούν σε μεγάλη κλίματα απαντήσεις, κλίμακα απαντήσεις και μάλιστα μακροπρόθεσμα. Μια στρατηγική λοιπόν που έχει θεμελιώδη σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είναι και ιστορικέ πολιτικέ, αλλά και πολιτισμικέ οι πολιτισμικοί δεσμοί που μα ενώνουν με τα κράτη αυτά. Αλλά και ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετανάστευση, την τρομοκρατία, την ανεργία των νέων, την κλιματική αλλαγή μα απασχολούν. Είναι στην Ευρώπη που πολλοί από τους νέους που κατέβηκαν στους δρόμους προσέβλεπαν περιμένοντας ε, περισσότερη δημοκρατία και πρόοδο και που η Ευρώπη έπρεπε να ενθαρρύνει δίνοντας κίνητρα αλλά με τα χρόνια και με την ανάδειξη της, διαρκούς, της διεθνούς τρομοκρατίας με το ίσις αλλά και μετά των μεταναστευτικών ροών. Αυτή η Ευρώπη λοιπόν στην οποία προσέβλεπαν περιορίστηκε στο να εξετάσει την σταθεροποίηση και την αποτροπή των μεταναστευτικών ροών μέσα από την πολιτική γειτονία του 2015 και μετά. Έτσι λοιπόν δεν επηρεάζει την περιοχή αυτή η Ευρώπη προς το καλύτερο, ούτε βελτιώνει τις συνθήκες ε, διαβίωσης των ε, πολιτών τους. Αντιθέτως έχουμε περιοριστεί στο να υποστηρίξουμε αυταρχικά καθεστώτα κατά τρόπο που δεν διαφέρει πολύ από το όσα κάνουμε στο παρελθόν. Δηλαδή κλείνουμε το μάτι σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θεμελιωδών ελευθεριών προκειμένου να μην έχουμε τρομοκρατία και μετανάστευση ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε τις θεμελιώδεις αξίες μας. Το μήνυμα που θέλω να αποστείλω με την έκθεσή μου είναι ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό. Ιδάλλως μόνο θα επαναλάβουμε τα προβλήματα του παρελθόντος και ακόμα και αν Έχουμε ε, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις του εις του 2011. Πρόκειται για μια ιστορία η οποία δεν μπορεί να τελειώσει σύντομα. Πρέπει να ε, οδηγήσει όμως μακροπρόθεσμα στην ειρήνη και την ασφάλεια ε, μια στρατηγική γενικότερη σφαιρική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπέβαλε και η κυρία Μογκερίνη το 2016 με μια έννοια κλειδί που είναι η ανθεκτικότητα των κρατών και των κοινωνιών των κρατών αυτών ε, με τα οποία έχουμε στενότερες σχέσει, των κρατών αυτών τη περιοχή. Και αυτό σημαίνει προοπτικέ ρεαλισμού, αλλά και αναγνώριση των αξιών μα. Η ανθεκτικότητα όμως δεν σημαίνει ταυτόχρονα σταθερότητα και συνέχιση της λειτουργίας των καθεστώτων αυτών, γιατί ένα αυταρχικό status quo αντιθέτως ε, αποτελεί αποσταθεροποιητικό παράγοντα, καθώς οδηγεί και σε διαφθορά, εγκληματικότητα, αποκλεισμό από την κοινωνία και ριζοσπαστικοποίηση. Άρα δεν είναι αυτό το κλειδί. Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε μια ρεαλιστική και θαραλέα προσέγγιση στην εργασία με τα κράτη-μέλη, με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του ρόλου της κοινωνίας των πολιτών, της, ε, της ανάδειξης των ικανοτήτων των νέων, και ταυτόχρονα αφήνοντας κατά μέρο τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα να κοιτάξουμε με κοινό βλέμμα τα κράτη αυτά. Τα κράτη αυτά που έχουν απογοητευτεί από την Ευρώπη και μπορεί να στρέψουν αλλού το βλέμμα, αλλού όπου οι αξίες μας, όπως άλλωστε έχει επισημανθεί και σε, θεμελι... σε θεσμικό επίπεδο από το χάρτη, ε, δεν γίνονται σεβαστές οι αρχές αυτές και οι αξίες, οι θεμελιώδεις αρχές και τα δικαιώματα δηλαδή η συμμετοχή των νέων στις διαδικασίες για τη λήψη των αποφάσεων θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά τρόπο που να τους επιτρέπεται η συμμετοχή τους στην κοινωνία, η ε, καταγραφή των θέσεων αυτών των ανθρώπων που ζουν σε αυτές τις κοινωνίες. Προτείνουμε συγκεκριμένα μέτρα για την υποστήριξη ισχυρότερης ε, πολιτικής και οικονομικής, κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Εδώ έχουμε τις τροπολογίες τώρα που έχω καταθέσει μια σειρά τροπολογιών για να συμπληρωθεί το κείμενο με δεδομένο ότι έπρεπε στην πρώτη εκδοχή του κειμένου να περιοριστώ στο αυστηρό, στα αυστηρά όρια του, που προβλέπονται ως προς τον αριθμό χαρακτήρων. Έχω βέβαια τις προτάσεις των συναδέλφων που θα ήθελα να δω. Είμαι αισιόδοξη ότι θα καταλήξουμε σε συμβαστικές τροπολογίες την επόμενη εβδομάδα πολύ εύκολα, χωρίς δυσκολίες, εν και της ψηφοφορίας των... Ε, Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τους και οδησηγητές ή τους αναπληρωτές τους. Ο κύριος Μπροκ αποουσιάζει, ο κύριος Ντανζό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον εισηγητή. Κατέθεσα τροπολογίες και ουσίες και τύπου διαδικαστικές εγώ θέλω να μιλούμε γενικώ στο πληθυντικό για τις αραβικές ανοίξεις, όχι μόνο στον ελληνικό, γιατί ιστορικά ε, ήταν διαφορετικές οι φάσεις ε, στις διάφορες χώρες. Και η κατάσταση είναι ανομοιογενής. Και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει έναν απολογισμό και να εφαρμόσει μια πιο συνεκτική ενωπημένη στρατηγική. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ε, έχουμε επίγνωση της ε, διαφορετικής κατάστασης που επικρατεί και της μεγάλης που υπάρχει μεταξύ των διαφορών χωρών. Γενικώ συμφωνώ με τους προσανατολισμούς της έκθεσης και κυρίως ε, στο ότι δυστυχώς ε, οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ήταν δυσανάλογες ή μάλλον δεν ανταποκρίνονταν στο αποτέλεσμα και στην προβολή αυτών των προσπαθειών λόγω της έλλειψης συνοχής που υπάρχει μεταξύ των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιμέρους πολιτικών των κρατών μελών για την περιοχή αυτή. Γι' αυτό δεν έγινε αρκετά ορατή η μεγάλη μας προσπάθεια. Και σίγουρα η περιοχή αυτή έχει στρατηγική σημασία για μα ε, τη ε, Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Πολύ περισσότερο σημαντική για μα από ότι για οποιοδήποτε άλλο εταίρο. Και θα πρέπει λοιπόν να τη δώσουμε την αξία που, ε, που δικαιούται, που τη αναλογεί. Και μπορεί να φαίνεται παράδοξο, αλλά δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις ό,τι αφορά το, την επιρροή που μπορούμε να ασκήσουμε και τη βαρύτητα. Και ναι, μεν έχουμε την εύλογη επιθυμία να επηρεάσουμε τη μεταβατική διαδικασία αυτών των χωρών, αλλά να αποφύγουμε να δώσουμε την αίσθηση μιας ε, επέμβασης, μιας παρέμβασης που θα αποκρουστεί από τις χώρες αυτές ε, ως ανεπιθύμητη. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε την ισορροπία. από τη μια να είμαστε δραστήριοι και να ενισχύσουμε την ε, επιρροή μας στην περιοχή, αλλά αποφεύγοντας μια αίσθηση ότι παρεμβαίνουμε κάτι που θα δημιουργήσει σε τα, στα αντίθετα και τελείως ανεπιθύμητα αποτελέσματα. Επίσης, πολλές φορές δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα και έμφαση στη σταθερότητα και στην ασφάλεια, βραχυπρόθεσμα, πρόθεσμα, εις βάρος μερικές φορές του μακροπρόθεσμου οράματος που χρειάζεται. Θα πρέπει επίσης την ανάγκη της ασφάλειας και της σταθερότητα να τη συνδυάσουμε με το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι πολύ σημαντική πρόκληση. Και συμφωνώ με τον εισηγητή ότι μερικές φορές δίνουμε υπερβολική έμφαση στη βραχυπρόθεσμη ασφάλεια, αλλά Α μην ξεχνούμε ότι οι προκλήσει ασφάλεια που αντιμετωπίζουν οι χώρε αυτέ είναι τεράστιε και λογικό είναι να λαμβάνονται υπόψη κατά προτεραιότητα στο μελλοντικό μα προσανατολισμό. Ευχαριστώ κύριο και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι δεδομένη τη μεγάλη ε, γεωγραφική εμβέλεια αυτών των περιοχών Μέση Ανατολή και Βορείου Αφρική και μάλιστα 8 χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη, είναι δύσκολο ε, και πολύ απαιτητικό το να καλύπτουμε με μια νέα προσέγγιση όλη την περιοχή και την ομοιομορφία της. Πάντως παρόλα αυτά είναι πολύ σημαντική η περιοχή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σίγουρα η ομάδα μου θα καταθέσει σημαντικές τροπολογίες και πολλές. Η μία φορά το θέμα της σταθερότητας στην περιοχή που είναι υπαριθμόν ένα προτεραιότητά μας αλλά ταυτόχρονα θέλουμε να ενθαρρύνουμε και να βοηθήσουμε ε, τις χώρες αυτές ε, ε, στον εκδημοκρατισμό τους και στην ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ανθρωπίνων ελευθεριών. Και θα πρέπει φυσικά να τις επιβραβεύουμε γι' αυτό, αλλά πρώτα απ' όλα οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να προσβλέπουν σε τέτοιες, σε ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να μην επιβάλλουμε εμείς αυτές τις απαιτήσει. Και από άποψη εξωτερικής πολιτικής θα πρέπει να συνεργαστούμε, να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία, ε, την ενίσχυση της ασφάλειας κατά της τρομοκρατίας και την ανάγκη της ε, πάταξης της διαφθοράς και της καταπολέμησης του εγκλήματος ε, και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και να αποφύγουμε επανάληψη ε, της κατάστασης του 2015 στα πλαίσια της μεταναστευτικής κρίσης και δεδομένων των πολλαπλών διακλαδώσεων που έχει αυτό το φαινόμενο θα επηρεάσει και τις ε, τοπικές μας, τις εχώριες μας πολιτικές. Στην περίπτωση, για παράδειγμα, του Brexit, ε, είχαμε πολύ ατυχή αφήσει στα πλαίσια της εκστρατείας για την αποχώρηση. Ε, Λέγοντα ότι η συμμετοχή μας, η ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας εμπόδισε να αποτρέψουμε ε, τη μεταναστευτική κρίση και να μην ξεχνούμε και το, τη μεγάλη απώλεια ανθρώπινων ζώων. Ε, θα καταθέσουμε, όπως είπα, τροπολογίες. Πάντως, γενικώ συμφωνούμε με την έκθεση, την κρίνουμε θετική και ευχαριστούμε τον κύριο Μπενιφέη για το σχέδιο που κατέθεσε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Τάνοκ. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω αγγλικά. Εγώ στηρίζω τη γενική προσέγγιση του εισηγητή γιατί θα πρέπει να κάνουμε μία επικριτική, αν θέλετε, αξιολόγηση της νέας στρατηγικής για την περιοχή αυτή. Και να σας πω επίσης πως στηρίζω την εξής άποψη υπερβολική σημασία δίνουμε στη σταθερότητα. Υπάρχει αυτή η ιδεολογία της σταθερότητας, όπως λέει ο εισηγητής. Τι σημαίνει αυτό. Υπάρχουν και άλλες προτεραιότητες, οι οποίες έχουν πάρει ε, δεύτερο ρόλο. Για παράδειγμα, και δημοκρατισμός, ανθρώπινα δικαιώματα και η κατάσταση στην περιοχή, κοινωνικο-οικονομικές ε, διαστάσεις, ανισότητα. Και έχουμε και μια άλλη συνέπεια στην πολιτική που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την περιοχή με βάκι αυτό είναι το ότι μπορεί να έχουμε μία προσέγγιση ε, στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά τα κράτη-μέλη έχουν τις δικές τους προτεραιότητες και τους δικούς τους στόχους. Και πιο συγκεκριμένα για κράτη τα οποία έχουν ιστορικούς δεσμούς με κάποια κράτη-μέλη και πολλές φορές αυτές οι στρατηγικές δεν ε, είναι... δεν συνδυάζονται μεταξύ τους. Η Αραβική Άνοιξη, οι πολλές περιπτώσεις Αραβικής Άνοιξης, κρύβουν τα προβλήματα αυτών των κοινωνιών ήταν ένα αίτημα για επέκταση ελευθερίας, αλλά η πραγματικότητα σήμερα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που φανταζόμασταν. Στις περισσότερες από τις χώρες αυτές έχουμε συνεχιζόμενα υψηλή διαφθορά, ε, έλλειψη λογοθοσίας, νεποτισμό, η κατάσταση με τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι κρίσιμη. Σε πολλές από αυτές τις χώρες και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να προκρίνουν τη στήριξη στα ανθρώπινα δικαιώματα σε όσους στηρίζουν αυτά στην κοινωνία των πολιτών. Έχουμε ένα πολύ ψηλό επίπεδο φτώχειας, ανισότητας. Δεν υπάρχουν ευκαιρίες για τους νέους. Και συνήθως η αντιτρομοκρατία και η νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο χρησιμοποιούνται ως τρόπους για να κατασταλεί οποιαδήποτε αντίρρηση και για να πιεστούν όσοι υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και η απάντηση στους πρόσφυγες και στις μετανάστες και στις ροές αυτές βασίζονται υπερβολικά ε, στις, ε, στα σώματα ασφαλείας και στην πτυχή ασφάλειας της πρόκλησης αυτής αφήνοντας στην άκρη την πιο ανθρώπινη απόκριση στο θέμα αυτό. Θα κλείσω λέγοντας πως εμείς υποβάλαμε 20 τροπολογίες και θα ήθελα να υπογραμμίσω μία από αυτές. Η περιοχή αυτή είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που προτείνω είναι να έχουμε εντολή για ειδικό ε, απεσταλμένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Νότια Μεσόγειο έτσι ώστε η πολιτική αυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή αυτή να είναι πιο ορατή και να ενισχυθεί από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σολέ εκ μέρους του κυρίου Κούλογλου, ο οποίος δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα, ε, θα σας διαβάσω ένα σημείωμα Ευχαριστώ τον κύριο Μπενιφέ ε, για τη δουλειά του που έχει πολλά στοιχεία θετικά στα οποία όμως μπορούμε να προσθέσουμε πολλά. 8 χρόνια μετά την Αραβική Άνοιξη, οι κυβερνήσεις εκεί εξακολουθούν να επιτίθονται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχουμε διδακτορικά καθεστώτα τα οποία παραμένουν με νέες κυβερνήσεις που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Όσοι απαιτούν μια πιο δίκαιη κοινωνία ε, πιέζονται και οι κοινωνίες αυτές έχουν τεράστια κοινωνική και οικονομική κρίση που οδήγησε στις διαμαρτυρίες του 2011 και που εξακολουθούν να δημιουργούν τέτοιου είδους διαμαρτυρίες. Έχουν τα επίπεδα ανεργίας που είναι τα υψηλότερα στον κόσμο, οι περικοπές, οι φόροι, τα βασικά προϊόντα και τιμές αυτών ήταν κάποιοι από τους λόγους που οδήγησαν στις διαδηλώσεις του 2011 και βρίσκονται πίσω και από τις νέες διαδηλώσεις που γίνονται. Θα πρέπει με ενεργητικό τρόπο να καταδικάσουμε το εμπόριο όπλων ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κάποιες από τις χώρες εκεί και ζητάμε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να επιβάλλει εμπάργο όπλων ε, κατά της Σαουδικής ε, Αραβίας λόγω της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου από τη χώρα αυτή. Μας ανησυχεί επίσης το γεγονός πως οι δικτατορίες στην περιοχή αυτή στηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ρόλο που ε, παίζουν οι ε, δυτικές παρεμβάσεις στην όξυνση των σειράξεων στην περιοχή. Οι πρόσφυγες και οι μετανάστες στην περιοχή αυτή ε, υποφέρουν, πολλοί έχουν βασανιστεί, τους έχουν εκμεταλλευτεί, τους έχουν βασανίσει, τους έχουν εκμεταλλευτεί σεξουαλικά η μάχη κατά της ε, τρομοκρατίας, της ε, ε, λαθρομετανάστευσης και της βίας δεν θα πρέπει να βασίζεται στην καταπίεση των ανθρωπινικών δημάτων στην περιοχή. Οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη λύση θα πρέπει να λάβει υπόψη την φτώχεια, την αστάθεια χώρες αυτές που είναι οι ρίζες των προβλημάτων και τα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών των λαών. Ελπίζω με τους υπόλοιπους σκιώδες να συνεργαστούμε θαυμάσια. Και αφού σας διάβασα τα όσα ήθελε να πει ο κύριος Στέλιος Κούλογλου. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρόκ. Äh, ναι, ευχαριστώ για την ευκαιρία να πω και εγώ κάτι εκ μέρους ομάδας μου αλλά και σε όρους ε, προσωπικούς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα σημαντικό ειδικό βάρος, αλλά δεν το έχει αξιοποιήσει κυρίως την πολιτική για την Αφρική. Χρειάζεται λοιπόν μια ιδιαίτερη ε, τοποθέτηση. Μετά τις αραβικές ανοίξεις, στην αραβική άνοιξη, εξελίχθηκαν διαφορετικά τα πράγματα στην κάθε χώρα. Και βλέπουμε για την Τινησία, παραδείγματι, που αποτελεί μια γενικά θετική εξέλιξη και το Μαρόκο που δεν έχουν πάει όλα τόσο στραβά, γενικά να πηγαίνουν χειρότερα τα πράγματα στις χώρες αυτές. Πρέπει λοιπόν να αναπτύξει περισσότερη οικονομική δραστηριότητα η περιοχή, αλλά και πολιτική ανθεκτικότητα. Και ένα ζήτημα βέβαια είναι το εμπόριο μεταξύ των κρατών αυτών. Οι δομές παραμένουν απεικιοκρατικές. περνούν ε, για τις σχέσεις τους χώρες αυτές μέσα από τις ε, παλές απεικιοκρατικές δυνάμεις και δεν έχουν μεταξύ τους επαφή. Ούτε απευθείας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ θα μπορούσε αυτό να βοηθήσει μια σαφέστερη οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικά την περιοχή. Θέλουμε και ελπίζουμε τα κράτη αυτά που είχαν ε, δικτατορίες αλλά που δεν είχαν πολύ συχνά ενελακτικές διεξόδους. Βλέπουμε παραδείγματι προς τα που τίνει η Αίγυπτος. Δεν μπορούμε όμως να λησμονούμε ποια ήταν η εναλλακτική. Καθόλου καλή και αυτή με την ε, μουσουλμανική αδελφότητα. Και εδώ, χωρίς να θέλω να καταδείξω κάποιον συγκεκριμένο υπέτειο, γιατί όλοι έχουμε συνυπευθυνότητα, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να δούμε και την πολιτική της Κίνας στην Αφρική και την διατάραξη των ειρηνευτικών προσπαθειών από πλευράς της Ρωσίας που ενθαρρύνει τις εμπόλεμες σειράξεις. Και έτσι κύριε Πρόεδρε, εγώ θα έβλεπα ότι υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τα κράτη. Και όχι η ίδια. Αυτό θεωρώ ότι θα ήταν ο καλύτερος δρόμος. Και νομίζω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε να βοηθήσουμε να σταθεί αυτή η περιοχή στα πόδια της. Είναι προς το συμφέρον όλων μας. Να είναι σταθερή αυτή η περιοχή της Μεσογείου, να προχωρήσει προς την ε, δημοκρατία, να προχωρήσει κοινωνικά, πολιτικά γιατί και για μας είναι σημαντικό να τη δούμε έτσι και για το θέμα της ε, μετανάστευσης βέβαια. Γιατί τα κράτη αυτά έχουν δυσκολία. Υποδέχονται μετανάστες από την ε, Μαύρη Αφρική με όλες τις φρικαλαιότητες που λαμβάνουν χώρα στο ταξίδι αυτών των ανθρώπων μέσα από τη Σαχάρα με βιασμούς, με παρανομές κρατήσεις. Μην ξεχνάμε ποιοι είναι αυτοί που το κάνουν. Πρέπει να τους αφοπλίσουμε και να επιτρέψουμε στις χώρες αυτές να αναπτυχθούν, να σταθούν στα πόδια τους, να προσφέρουν μια καλύτερη κατάσταση στους πολίτες τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπροκ. Το λόγο κύριε Λαλάν, τελευταία μας ομιλήτρια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μια και έφυγε η κυρία Φάουτμανς, που είναι και η σκιώδη για των Φιλελευθέρων για το θέμα αυτό, θα σας παρουσιάσω εγώ τα σχόλιά της για την έκθεση, για την εποχή μετά την Αραβική άνοιξη και ποια είναι η ακολουθητή απορία στην περιοχή Μέση Ανατολή και Βορειοαφρική. Η κυρία Φάουτμαν σε ευχαριστεί τον εισηγητή τον κύριο Μπενιφέ για την εξαιρετική έκθεση, το σχέδιο έκθεσή του, γιατί είναι άρτια και επικεντρώνεται στα κατάλληλα σημεία. Την ανάγκη δηλαδή να αναπτυχθεί νέα πολιτική για την περιοχή ΜΑΒΑ που θα συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη οικονομική και πολιτική σταθερότητα των χωρών τη Μέση Ανατολή και Βορειοαφρική. Η κυρία Φάουτμαν, συσκιώδη συγγετρία, θα καταθέσει και τροπολογίε στην έκθεση Benifei, πιο σημαντικές είναι οι εξή. Έχουμε τη τελική σκέψη για την ενίσχυση της καταστολής ε, εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών σε πολλές χώρες ΜΑΒΑ. Πολλές ε, κοινοτικές χώρες συνεχίζουν ε, να εξάγουν τεχνολογίες επιτήρησης προς χώρες ΜΑΒΑ διευκολύνουν τη διαδικτυακή παρέμβαση και άρα και τις επιθέσεις προς ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στηρίζουμε τις βλέψεις των λαών των χώρων της Μέσης Ανατολής και της Βορειοαφρικής που είναι υπέρ δημοκρατικών ευήμερων κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς. Επίσης, η μακροπρόθεσμη ευημερία των χωρών αυτών συμβαδίζει με την προστασία των οικουμενικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη θέσπιση δημοκρατικών και διαφανών θεσμών που θα προστατεύουν τους πολίτες και τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Καταδικάζουμε τη χρήση ε, του επιχείρηματος της ασφάλειας ε, ή της αντιτρομοκρατίας σε κάποιες χώρες της περιοχής για, ως πρόσχημα για την καταστολή της ελευθερίας έκφρασης. Χαιρετίζουμε την ε, στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις χώρες αυτές και επαναλαμβάνουμε την ανάγκη να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να αντιμετωπίσουμε τα αίτια των συγκρούσεων. Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας για την πιθανή εργαλειοποίηση της, ευρωπαϊκής, της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση της μετανάστευσης. Επίσης, επικεντρωνόμαστε σε μια χώρα, κυρίως στη Συρία, καταδικάζουμε δρυμύτατα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έγιναν κατάφορα στη διάρκεια τη σύγκρουση μετά τι επανειλημμένε αποτυχίε ε, τη κατάπαυση των βιοπραγιών και των εχθροπραξιών και επισημαίνουμε την ανάγκη να βρεθεί μια βιώσιμη λύση ειρηνευτική. Επίσης δεν θα πρέπει ε, να εφαρμοστεί ατιμορρησία για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν στη Συρία. Ευχαριστώ κύριε Λαλόντ. Ελάχιστος χρόνος μας έχει μείνει και μας, έχω δύο ακόμη ομιλητέ. Τους θερμοπαρακαλώ να είναι πολύ λακωνικοί για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε εγκαίρως τη συνεδρίασή μας. Ο κύριος Ζιλμπερτράν καταρχήν που είναι σύμβουλος του αναπληρωτή διευθυντή για την περιοχή ΜΑΒΑ στην ΙΕΤ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί με την έκθεση αυτή παίρνετε μία απόσταση και προσπαθείτε να υιοθετήσετε μια πιο συγκροτημένη ε, άποψη για τις πολιτικές μας και πιο διαφθορετική και δεν επικεντρώνεστε μόνο στις οξύες κρίσεις. Η έκθεση που πραγματεύεται την εποχή μετά την Αραβική Άνοιξη επισημαίνει πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο. Είναι δύσκολο ακόμη και να κρίνουμε ε, το που η ιστορία θα ε, εξωθεί στις χώρες του ΜΑΒΑ. Ε, λίγα χρόνια έχουν περάσει ακόμη, μόνο 8. Σε 20-30 χρόνια θα έχουμε πολύ διαφορετική άποψη για το τι συνέβη ή δεν συνέβη στην περιοχή. Πάντως πολύ ε, εύστοχα η έκθεση επισημαίνει ότι δεν έχουμε καθόλου ούριο άνεμο στην περιοχή. Είναι πολύ αρνητικές για τη δημοκρατία παγκόσμια τάσεις. Υπάρχουν περίπλοκα θέματα, ασφάλεια, μετανάστευση, περίπλοκες τάσεις ακόμη και στις κοινωνίες των, των χωρών της ε- Μέσης Ανατολής και της Βορειοαφρικής, κάτι που καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από ότι στο πρόσφατο παρελθόν. Τώρα, εν συντομία, λαμβάνοντας υπόψη της ε, επικρίσης και την εικόνα που παρουσιάζει η έκθεση, θα ήθελα να πω ότι κάναμε κάποιες προσπάθειες για να παραμείνουμε προβλέψιμος εταίρος στην περιοχή. Και θεωρούμε ότι τη στιγμή που όλο και περισσότεροι παγκόσμιοι εταίροι γίνονται απρόβλεπτοι, είναι σημαντικό εμείς να είμαστε προβλέψιμοι και αυτό το χαιρετίζουν και οι εταίροι μας στις χώρες αυτές. Τα τελευταία χρόνια προσπαθήσαμε να στηρίξουμε τις χώρες Μέση Ανατολής και Βορειοαφρικής για να αντιμετωπίσουν τους περιφερειακούς κραδασμούς ιδιαίτερα την επαύριο των κρίσεων των γειτονικών τους χωρών. Για παράδειγμα, η αντίδραση στη Συριακή κρίση, στο Λίβανο, την Ιορδανία και το πώς στηρίξαμε αυτές τις χώρες για να αντιμετωπίσουν αυτή την έλλειψη σταθερότητας αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να ενισχύσουν τη δική τους σταθερότητα. Επίσης, προσπαθήσαμε να στηρίξουμε και την κοινωνία των πολιτών και τους ΜΚΟ για, και να κρατήσουμε τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα ανθρώπινα δικαιώματα ύψιστη προτεραιότητα. Και μάλιστα στις χώρες αυτές ε, βασική μας εταίροι είναι η κοινωνία των πολιτών, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, οι οργανώσεις νεολαίας που δραστηριοποιούνται υπέρ της δημοκρατίας και θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο των σχέσεών μας. Σε ό,τι αφορά την ανάληψη ευθύνης για την πολιτική της γειτονίας και από πλευράς εταίρων. Αυτή είναι μια σχετικά καινούρια αλλαγή στην πολιτική και είναι πολύ νωρί για να κρίνουμε τα αποτελέσματα, να τα αξιολογήσουμε. Το γεγονό ότι τώρα διαμορφώνουμε τι προτεραιότητε μα, αποκοινούμε του εταίρου μα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει στην επιλογή μόνο των σημείων που μα συμφέρουν, που μα βολεύουν. Και στο παρελθόν το πρόγραμμά μας ε, διαμορφώνονται κυρίως με βάση τις δικές μας προτεραιότητες, με γνώμονα τα δικά μας συμφέροντα και όχι με βάση κοινέ προτεραιότητες, κάτι που θα είναι η νέα πρόπτικη. Πάντως ε, σε όλες τις ε, προτεραιότητες που συμφωνήσαμε, η κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία είναι βασικό στοιχείο των προτεραιοτήτων. Βέβαια δεν ήταν καθόλου πάντα εύκολη διαδικασία με όλους τους εταίρους, αλλά σε αυτό επιμείναμε στις διαπραγματεύσεις τους τους τομείς. Και τέλος, η έκθεση πολύ στο, σωστά επισημαίνει το θέμα της νεολαίας και τη στήριξη που μπορούμε να προσφέρουμε σε οργανώσεις νεολαίας. Είναι ένα θέμα που προσέχουμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, όπως και η στήριξη των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, όπου μπορούμε φυσικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μίλλερ, λοιπόν, που είναι επικεφαλής ε, της Μονάδας για τη Μέση Ανατολή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε το λόγο για να σχολιάσω και εγώ την έκθεση αυτή. Ξέρετε και εσείς πως ξανακοιτάξαμε την πολιτική αυτή το 2015 και τότε αποφασίσαμε πως θέλουμε την σταθερότητα και την ανθεκτικότητα να την τοποθετήσουμε στην κορυφή των προτεραιοτήτων της πολιτικής γειτονίας. Και είπαμε, θα είμαστε λιγότερο περιγραφικοί σε αυτά που επιθυμούμε από τους συνεργάτες μας και τους εταίρους μας στα πλαίσια αυτής της πολιτικής και θέλουμε να έχουμε ε, σταθερότητα κοινωνική, οικονομική και αναγνωρίζουμε πως αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις με τον εξυγχρονισμό όπου το κοινωνικό συμβόλαιο σε πολλές χώρες είναι αδύναμο, ανύπαρκτο και που χρειάζεται να ανασυγκροτηθεί. Και τα τελευταία 8 χρόνια από την Αραβική Άνοιξη θα δείτε πως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν ε, ε, επηρεάζουμε και ε, ευθυγραμμίζουμε τις δικές μας απαιτήσεις με αυτές των γειτόνων μας μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Και όπου ήμασταν αποφασιστικοί ε, και είχαμε κοινού στόχου ε, μαζί με του γειτονέ μα, ήμασταν αποτελεσματικοί. Και του βοηθήσαμε με κοινού στόχου στην πολιτική μεταρρυθμίσεων, δίνοντα την ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί μα. Αυτή η διαφοροποιημένη προσέγγιση ήταν ζωτική σημασία για να αναζωπηρωθούν οι σχέσει μα με τι χώρε ε, στα πλαίσια τη πολιτική γειτονία. να εστιάσουμε εκεί που μπορούμε να φέρουμε τη διαφορά και η υπηρεσία εξωτερική δράση έχει ήδη σχολιάσει τις ε, διαπραγματεύσεις των προτεραιοτήτων εταιρική σχέσης που είναι πολύ σημαντικές στα πλαίσια αυτά. Στις συζητήσεις με τους εταίρους μας ήμασταν σαφείς. Ε, κοινέ αξίες και κοινά συμφέροντα. Είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος και δεν μπορούν αυτά να επιτευχθούν όταν δεν υπάρχουν ε, εναλλακτικέ για την κρατική, τον κρατικό έλεγχο της οικονομίας και για την ευημερία της κοινωνίας των πολιτών. Πρέπει έχουμε ε, θεσμούς που λογοδοτούν, χρηστή διαχείριση και δικαιώματα για όλου. Αυτά είναι ζητική σημασία όπω επίση και ευκαιρίε για την νεολαία. Και βρήκαμε πως η οικονομική μας ε, συνεισφορά στην περιοχή θα πρέπει να παραδίδεται με ένα βελτιωμένο τρόπο. Βέβαια, όταν δεν υπάρχει πολιτική βούληση, εμείς δεν μπορούμε αυτή να την προσφέρουμε. Και δεύτερον, πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ ε, των κινήτρων που δίνουμε, αλλά και της προβλεψιμότητας των οικονομικών, ροών που είναι απαραίτητες για μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, για την πολιτική βούληση. Θα πω το εξή. Εμείς συνεργαστήκαμε εντατικότατα ε, με το Ευρωπαϊκό Όργανο για Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και έχουμε ε, ενισχύσει την εργασία μας με το Ίδρυμα ε, το σχετικό για την περιοχή της, ε, των χωρών νοτίους γειτονίας και δεν έχουμε βρει έναν τρόπο να συνεργαζόμαστε με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις εύκολα. Πάντως έχουμε πει πως είναι πολύ αποτελεσματικά τα όργανα που χρησιμοποίησαμε και ο μηχανισμός παρόλη την κριτική από το ελεγκτικό συνέδριο και ε, για την συνοχή, την ε, να σας πω πως στη Νότια Ευρώπη ήταν πάρα πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα εκεί, αλλά δυστυχώς έχουμε το πρόβλημα της, ε, του μη συντονισμού με το όσα κάνουν τα Ταμεία Συνοχής στα κράτη-μέλη. Εκεί έχουμε και μια παρατήρηση στην έκθεση. Τώρα, για τα συμβουλευτικά ε, όργανα τα οποία προβλέπονται στην έκθεση, εμείς δεν θεωρούμε πως είναι κάτι το εύχριστο. Υπάρχει ο, κόσμος, υπάρχει ο κίνδυνος να συζητάμε με αυτούς οι οποίοι μόνο μαζί μας συμφωνούν. Ε, και αποκλειστικά με αυτού. Οπότε είπαμε, μη κυβερνητικέ οργανώσει, κοινωνία των πολιτών, οι εκπρόσωποι θα πρέπει να μιλάνε με τι εθνικέ διοικήσει, έτσι ώστε από την αρχή τη χάραξη πολιτική να συμμετέχουν. Εμεί, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να του διευκολύνουμε. Αυτή ήταν η εμπειρία μου από τις της Ευρωπαϊκή Ένωση εκτό και μπορούμε να σχεδιάσουμε παρεμβάσει, οι οποίε δίνουν έναν ρόλο παρακολούθηση στην κοινωνία των πολιτών. Αλλά εμεί δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε αυτή τη σχέση που θα υπάρχει μεταξύ τη κοινωνία των πολιτών και των κυβερνητικών αρχών. Θα πρέπει επικοδομητικά αυτοί να συνεχιστούν μεταξύ τους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω πως για τις τροπολογίες έχουμε μέχρι 17 Ιανουαρίου έχουμε λάβει 265 ήδη. Λάβατε υπόψη πως ε, 20 Μαρτίου του 2018 το Διευθυνμένο Προεδρείο είπε πως τροπολογίες μπορούν να καταθέτουν μόνο για τις χώρες που είναι ε, χώρες της ε, Αραβικής Άνοιξης, δηλαδή νότια Μεσογείου. Αύριο ακρόαση για το θέμα αυτό, από τις 2.30 μέχρι τις 3.30. Ωραία λοιπόν, στα γρήγορα να περάσουμε στο σημείο 14, να σας υπενθυμίσω όπως είπε ο κύριος Μακάλης, έχουμε πάρα πολλά σημεία και γι' αυτό σας συζητώ να είστε πολύ σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Τώρα θα δούμε το σχέδιο σύστασης για τη Συμφωνία σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανδόρας, ε, Μονακό και Σαν Μαρίνο και Άγιο Μαρίνο. Τα τρία αυτά ευρωπαϊκά κρέτη, το θέμα είναι υποδιαπραγμάτευση και το σχέδιο σύστασης έχει ως στόχο να ορίσουμε τα βασικά σημεία και να περιγράψει ανησυχίες του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Λόπες Αγγελάρη έχει το λόγο μια κοινή Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, με μεγάλη χαρά παρουσιάζω το σχέδιο αυτό έκθεσης για τη σύσταση η Επιτροπή ΑΦΕΤ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ανέλαβε δυνάμει της συνθήκης Λισαβόνα στην εξουσία να χορηγεί συνένεση σύμφωνη γνώμη ή καλύτερα να χαράζει το δρόμο για τη σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου και τελική έγκριση διεθνού συμφωνία για τη θέση, ενόψη θέση ενισχύση τη διεθνή συμφωνία λοιπόν μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση ή οδήποτε τρίτου μέρους. Εδώ έχουμε λοιπόν μια συμφωνία σύνδεσης μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, της Ανδόρας, του Μονακό και του Αγίου Μαρίνου, τριών μικρών κρατών, μικροκρατών θα μπορούσα να πω, και δεν θέλω να καταστήσω σαφές εξ αρχής προσεφής της συμφωνία στηρίζεται στην επικρατούσα διαπραγματευτική εντολή που χορήγησε το Συμβούλιο στην Επιτροπή για να διαπραγματευτεί εκ μέρους του. Και το λέω αυτό γιατί είναι σημαντικό για να προσδιορίσουμε το πεδίο της συζήτηση από εδώ και μπρο. Εδώ μιλούμε για τη συμμετοχή τριών μικρών ακόμη κρατών, μικροκρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ιστορική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από τις ε, τέσσερις ε, ελευθερίες οι οποίες εγκαθιδρύονται και για τις χώρες αυτές με την ενσωμάτωση του κοινοτικού κεκτημένου. Το λέω αυτό διότι είναι προφανές. ότι πάντα ε, όταν έρχεται η ώρα να συστήσουμε οικονομικά συστήματα για τα τρία αυτά μικρά κράτη παρα... Ε, ε, παρασυρώμαστε σε κλεισές κοινοτοπίε. κοινοτοπίες. Εγώ είμαι διτεθειμένος να αγωνιστώ πάντα και για την ε... διαφάνεια τη φορολογική, για την καταπολέμηση της φοροαπάτης, φοροαποφυγής, νομοποίησης παρανομών εσόδων. Έχω αφιερώσω όλη μου τη ζωή και τη αδρομία στο πεδίο αυτό. Και ως υπουργό ε, δικαιοσύνης της Ισπανίας στο παρελθόν, είχα την ευθύνη της ανάπτυξης των ε, εργασιών του γραφείου του ε, εισαγγελέα του, του κράτους. Ωστόσο, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε τέτοια θέματα, έχουμε να κάνουμε τις ελευθερίες. Τα θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου και του ΕΚΟΦΗΝ, αλλά και πέραν αυτών, το όσα ε, το Συμβούλιο της, της Ευρώπης, μας λένε με τις εκθέσεις τους πως οι χώρες αυτές έχουν απόλυτη συμμόρφωση και υποταγή όσον αφορά τη διαφάνεια στη φορολογία και την νομιμοποίηση παρανομών εσόδων με τους κανόνες. Άρα λοιπόν ε, μπορεί κανείς να αναφέρεται σε κάποιες κακές ημέρες, ε, εποχές στο παρελθόν, τις άρεστες καταστάσεις που όμως τώρα έχουν αλλάξει και ανοίγει ένα νέο πλαίσιο πολιτικών σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών αυτών. Ένα μέλλον όπου αυτές οι χώρες έχουν αναπτύξει ε, πρότυπα κοινά έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορούν να καταλάβουν το χώρο τους ως ισότιμοι εταίροι. Η Ανδόρα, το Μονακό και, το, και ο Άγιος Μαρίνος έχουν ε, πραγματοποιήσει σημαντικέ μεταρρυθμίσεις και ρυθμιστικές αναθεωρήσεις, ιδιαίτερα σχέση με τον κανονισμό, το σχετικό με την τραπεζική δραστηριότητα και τα χρηματοπιστωτικά, αλλά και την καταπίεση της νομοποίησης παρανόμων εξόδων και ε, του οικονομικού εγκλήματος ίσως αργότερα ο κ. Μόρτον που ήταν ο υπεύθυνο διαπραγματεύτη εκ μέρου τη Επιτροπή, να έχει την ευκαιρία να μα διευκρινίσει τα σημεία αυτά. Αλλά για την ουσία. Ξεκινούμε με το άρθρο 11, δήλωση από την συνθήκη τη Λισαβονά, που λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδιαίτερω υπόψη ε, προβλήματα που απορρέουν από το μικρό μέγεθο ορισμένων κρατών. Τρία κράτη λοιπόν, τα οποία είναι όντως πολύ μικρά, βέβαια είναι ευρωπαϊκά ως προς τη φύση τους και τη γεωγραφία τους. Ε, εδώ έχουμε να κάνουμε σχέση μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας, Γαλλίας-Ιταλίας, στην περίπτωση του Μονακό και εσωτερικό της Ιταλίας στην περίπτωση του. Παρακαλώ αν έχετε την καλοσύνη να ολοκληρώνετε. Μα ένα λεπτό. Άκουσα τόση ώρα να μιλάει η Κομισιόν. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Ε, σας είπα να ολοκληρώσετε. Ήδη μιλήσετε πέντε λεπτά. Το πω. Μα όχι, θέλω να τα πω. Η ιδέα λοιπόν εδώ είναι να αποστείλουμε ένα θετικό μήνυμα σε όλους τους εμπλικόμενους ε, φορείς και τα μέρη, να τα ενθαρρύνουμε έχουμε την ευκαιρία να επιδείξουμε ευελιξία ε, και επιτυχία στην έκβαση των συνομιλιών. Ετοιμάζουμε το σχέδιο μετά την επίσκεψη στις τρεις αυτές χώρες για να περιγράψουμε σωστά την κατάσταση και θεωρώ ότι θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Θα ήταν αποτυχία και για τις δύο πλευρές της ε, όχι μόνο τα μικροκράτη αυτά, αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να μην στεφθεί με επιτυχία η διαπραγμάτευση. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, πρέπει να αντιληφθούμε ότι η εσωτερικά και αγορά και τέσσερι ελευθερίες δεν κινδυνεύουν από τη Συμφωνία Σύνδεσης. Άρα ευελιξία στην ενσωμάτωση του κεκτημένου θα πρέπει να είναι δεδομένη. Και πρέπει να εξασφαλίσουμε εταιρική σχέση με τις τρεις αυτές χώρες, αλλά χωριστά με την καθεμία γιατί δεν έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά όλες μικρές χώρες μεν, αλλά με διαφορές μεταξύ τους. Ε, για την ε, Ανδόρα, παραδείγματα, έχει πολύ μεγάλη σημασία η διαφύλαξη του τομέα των, ε, των προϊόντων καπνού. Όχι, όχι, θα συνεχίσω. Λοιπόν, το ίδιο για τον Άγιο Μαρίνο, εξαγωγέ και για το Μονακό, η κύρια ανησυχία που εκφράζει είναι η διαφύλαξη της δυνατότητας να διατηρηθούν οι κάτοικοι που γράφονται εκεί, ξέροντας ότι οι μόνιμοι κάτοικοι, οι πραγματικοί κάτοικοι είναι ε, πολύ λίγοι σε σχέση με αυτούς που δηλώνουν διαμονή εκεί, τους αλλοδαπούς ε, που έχουν διαμονή. Γι' αυτό λοιπόν ε, πρέπει να διαφυλαχθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των χωρών αυτών. 50 ήταν οι τροπολογίες, έχω λάβει υπόψη, με κύρια ιδέα να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία 4 Φεβρουαρίου στην ΑΦΕΤ και στην πρώτη Ολομέλεια το Φεβρουάριο. Ε, εσείς να με συμπαθάτε, αλλά έχουμε ένα ακόμη σημείο και δεν θα έχουμε διερμηνία. Αλλιώς θα πρέπει να περιορίσω τους υπόλοιπους ομιλητές στο δίλεπτο, ενώ εσείς μιλήσατε 9 λεπτά. Εκτός μικροφώνου, ο κύριος Λόπες Εν πάση περιπτώσει, δεν ισχύει αυτό που λέτε. Μιλήσατε 4 λεπτά και... Θα δώσω τώρα το λόγο στους και Σιωπή παρακαλώ. Η κυρία Ζόφκο. Δύο λεπτά παρακαλώ οι σκιοδησηγητές γιατί οι διερμηνείς ε, θα πρέπει να φύγουν. Σας ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συναδελφοί, ως και ηγετρία για τη σύσταση προς το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ανδόρας Μονακό και Αγίου Μαρίνου, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και το έργο του. Χαιρετίζω τα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για τις διαπραγματεύσεις με τις τρεις χώρες. Είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και προς το συμφέρον των τριών χωρών να ενισχυθούν οι σχέσεις μας και να αξιοποιήσουμε τις κοινέ μας πολιτικές, πολιτιστικές και άλλες αξίες για να οδεύσουμε προς ένα αρμονικό κοινό μέλλον. Η εξασφάλιση της πρόσβασης στην ενιαία αγορά και η εθάρρυνση της εφαρμογής των τεσσάρων θεμελιωδών ευθελειών θα οδηγήσει σε στενότερη συνεργασία με τις γειτονικές αυτές χώρες βάσει του κοινοτικού κεκτημένου, ε, κάτι που θα είναι μια αμοιβαία υποφελής κατάσταση δεδομένης της μικρής εδαφικής έκτασης και των τριών χωρών, είπα στην τροπολογία μου πόσο σημαντική είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου για να εφαρμοστεί η Συμφωνία Σύνδεσης με τις τρεις χώρες και να εξασφαλίσουμε μια συνεπή εφαρμογή και ερμηνεία του κοινωτικού κεκτημένου στις τρεις επιμέρους χώρες. Ε, επίσης, θα ήθελα να ε, υποστηρίξω τη συνέχιση της διαδικασίας και να ενθαρρύνω την άμεση ολοκλήρωση και διεκπαιρέωση της Συμφωνίας Σύνδεσης. Ευχαριστώ κυρία Σοφκό, κύριο και Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ επιγραμματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Λόπες Αγγιλάρ. Ήμουν πάντα ε, φίλος των μικροκρατών αυτών της Ευρώπης. Ε, στο ένα έχω οικογένεια, στο αλλά έχω πάει έχω φίλους στην Άνδρα, έχουν μια μοναδική ιστορία, έχουν μια ε, κοινή ιστορία και αξίες ε, που τα κάνουν πολύ ξεχωριστά, που θα πρέπει να διατηρηθούν και είναι ένα εξαιρετικό συμβιβασμό για να έρθουμε πιο κοντά μέσω αυτή τη επόμενη συμφωνία σύνδεση, ενισχύοντα τι ε, σχέσει που έχουμε, ε, συνεργασία τύπου Τελωνιακή Ένωση, ε, συμφωνία σύνδεση και για να πατάξουμε το οργανωμένο έγκλημα και την ε, το ξέπλυμα χρήματο. Βέβαια, για τις τέσσερι ελευθερίες πρέπει να έχουμε ένα περιορισμό τη ελευθερία μετακίνηση μετακίνησης, γιατί είναι πολύ μικρά κράτη και νομίζω πως είναι περίεργο που η χώρα μου που θα περάσει τον Brexit θέλει να σταματήσει την ελεύθερη κυκλοφορία των ανθρώπων εγώ δεν μπορώ να αντιμετωπίσω με συμπάθεια μια χώρα 65 εκατομμυρίων που ανισχύει για κάτι τέτοιο. Μετακινήσει τέτοιε μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, όμω τα μικροκράτη δεν μπορούν και γι' αυτό θα πρέπει να ε, το λάβουμε υπόψη μα αυτό, παροτρύνοντά του να έρθουν πιο κοντά μα και ελπίζουμε ε, πως στο μέλλον θα βρούμε και έναν τρόπο να γίνουν μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. με το δικό του ειδικό καθεστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Νάρτ έχει το λόγο. Το πρόβλημα δεν είναι η βιομηχανική παραγωγή του Αγίου Μαρίνου, της Ανδόρας ή του Μονακό αλίμονο. Το πρόβλημα είναι η χρηματοπιστωτική πλατφόρμα. Αυτά, αυτή είναι η χρηματοπιστωτικη πλατφορμα αυτη ειναι η κατασταση Και ας δούμε το εξή. Εγώ πιστεύω ότι το Άγιο Πνεύμα δεν έπεσε στο Μονακό, ούτε στον Άγιο Μαρίνο, ούτε στην Ανδόρα. Δεν τους ήρθε επιφύτηση. Η μεγάλη διαφορά του κατακεφαλήν εισοδήματο προέρχεται από τι προνομιακέ καταστάσει που ζουν. Γι αυτό, ε, άλλωστε και το Γεβραλτάρ είναι τρίτη, το τρίτο κατακεφαλήν εισόδημα στον κόσμο. Όχι επειδή είναι τόσο έξυπνοι κάτι κάτοικοι του Γεβραλτάρ, αλλά επειδή έχουν καταπληκτικέ χρηματοπιστωτικέ υπηρεσίε ε, και προσφέρουν σε σχέση με την Ισπανία, για παράδειγμα. Οπότε α έχουμε υπόψη αυτό το κρατούμενο, ότι η κατάσταση ε, των εδαφών αυτών δεν είναι κατάσταση κρατών απόρων, αλλά χωρών που έχουν κατακεφαλήν εισόδημα υψηλότερο από τι γειτονικέ χώρε, όχι λόγω των ικανοτήτων που έχουν οι κάτοικοι των χωρών αυτών, αλλά λόγω τη ιδιάζουσα θέση και των ιδιαίτερων προνομίων που απολαμβάνουν ε, και των, ε, της γητά τους προς άλλες χώρες που δεν εφαρμόζουν αντίστοιχα προνόμια. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να θελοτυφλούμε. Είχαμε σοβαρά, σοβαρότατα σκάνδαλα που παρεμποδίσαμε, αλλά αφού έγιναν τα σκάνδαλα, δηλαδή κατόπιν εορτής, δεν τα προλάβαμε, είναι σημαντικό λοιπόν, αν μιλούμε για εσωτερική αγορά, Α μην ξεχνούμε ότι δεν υπάρχει εσωτερική αγορά που δεν θα καλύπτει και τι χρηματοπιστωτικέ συναλλαγέ. Εδώ δεν μιλούμε για την παραγωγή του καπνού ποικιλία Ρόσλη στην Ανδώρα. Μιλούμε για άλλη κατάσταση, αυτή που αντιστοιχεί στην απόλυτη, ξεκάθαρη, διαφανή και πλήρη συνεργασία που θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ αυτών των χωρών, αυτών των κρατών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά το, το ξέπλυμα χρήματο και τη φοροδιαφυγή. Και υπάρχει και μια λειτουργία που είναι εξαιρετικά σημαντική. Ο εντοπισμός των πραγματικών δικαιούχων. Γιατί μόνο τους εικονικούς δικαιούχους γνωρίζουμε ή τους ε, ε, εικονικούς κατόχους ε, των αμύθιτων περιουσιών όχι τους πραγματικούς κυρίους. Και η μικρή έκταση δεν σημαίνει ε, ίσονο σημασία οικονομική δύναμη. Το αντίθετο, ειδικά για την περίπτωση αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Νάρτο. Κύριος ε, Γιόρντι, Τζόρντι έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Καταρχήν, συμφωνώ με τον εισηγητή ότι είναι σκόπιμο να βελτιώσουμε και να εμβαθύνουμε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα τρία αυτά μικροκράτη, την Ανδόρα, τον Άγιο Μαρίνο και τον Μονακό. Γιατί πρόκειται για ευρωπαϊκά εδάφη και το κοινό μας σημείο δεν είναι μόνο η γεωγραφία, αλλά και η ιστορία και οι κοινέ μας αξίες. Δεύτερο θέμα. Στις διαπραγματεύσεις ε, για τη Συμφωνία Σύνδεσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες αυτών των κρατών που έχουν φυσικά μια κρατικότητα και μακρά ιστορική πορεία, μακρόχρονη ιστορία, αλλά και κάποιες πολύ ιδιαίτερε συνθήκες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις ιδιαιτερότητες, όλες αυτές τις ιδιομορφίες των συγκεκριμένων χωρών. Και τρίτον, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι χώρες αυτές και την πρόοδο που σημείωσαν αυτά τα μικροκράτη λόγω γεωγραφική και πολιτιστική συγκίτας, εγώ είμαι περισσότερο εξοικειωμένο με την κατάσταση στην Ανδώρα. Έκανε τεράστιε προσπάθειε για να βελτιώσει την ομοθεσία τη για να έχει πιο διαφοροποιημένη οικονομία. Ταυτόχρονα όμω, ελπίζω αυτέ οι νέε σχέσει που θα έχουμε με τα τρία αυτά μικροκράτη να δώσει και ενάψματα στι τρει αυτέ χώρε να συνεχίσουν τι προσπάθειές του και να βελτιώσουν την κατάσταση στη φορολογία, για παράδειγμα, και στη διαφάνεια. Εκεί όντως έχει συντελεστεί πρόοδος, αλλά δεν αρκεί και θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες και σε αυτά τα τρία μικροκράτη, αλλά και εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι η Ανδώρα είναι η μοναδική χώρα του κόσμου που έχει τα καταλανικά ως επίσημη γλώσσα. Έχουμε τρεις χώρες μέλη στις οποίες ε, μιλούνται τα καταλανικά, αλλά δεν είναι επίσημη γλώσσα. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώ δεν μπορώ σήμερα να σα μιλήσω, είναι γενικώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μιλώ στα καταλανικά. Τέλο, ο κύριο Μάρτιν, επικεφαλή τη ε, Μονάδα για τη Δυτική Ευρώπη, παρακαλώ πολύ και εσεί να είστε σύντομο, γιατί μα έχει μείνει ένα σημείο ακόμα. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τα σχόλια που κάνατε. για το σχέδιο αυτοσύσταση που είναι πολύ σημαντικό για τις διαπραγματεύσεις. Είναι εδώ και τρία χρόνια που διαπραγματευόμαστε με αυτά τα τρία κράτη και είναι σημαντικό σήμερα να στείλουμε ένα στεναρό πολιτικό μήνυμα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να δείξουμε στις χώρες αυτές την πολιτική σημασία που δίνουμε στις διαπραγματεύσεις αυτές για τη συμμετοχή στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι τρεις χώρες είναι πολύ κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμεριζόνται τις αξίες μας. Σήμερα έχουν πρόσβαση που δεν είναι αρκετή για να δρέψουν τα πλονεκτήματα, τα πιθανά πλονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Εσωτερικής Αγοράς. Θέλουμε λοιπόν με τη συμφωνία να τους δώσουμε πρόσβαση, βέβαια με το δικαίωμα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται ε, μέσω του ε, ευρωπαϊκού κεκτημένου και των τεσσάρων ελευθεριών. Είναι μικρό το μέγεθος των χωρών αυτών και ίσως γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε ευέλικτοι, λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση άρθρου 8 της συνθήκης, κάτι το οποίο γίνεται, και αυτή η ευελιξία θα προσφερθεί όπου μπορούμε. Όμως θα πρέπει το κεκτημένο να ληφθεί υπόψη και να εφαρμοστεί και ως προς τις τέσσερις ελευθερίες χωρίς εξαίρεση για αυτές τις χώρες αυτές. Έχουμε και ένα μηχανισμό ελέγχου και παρακολούθησης που προβλέπεται από τη διαπραγμάτευση για το πολυμερές ε, ε τμήμα που διαπραγματοβόμαστε με αυτές τις χώρες και έχουμε ένα σύστημα που θα λαμβάνει υπόψη και τις αποφάσεις του ΔΕΚ και το ρόλο του ΔΕΚ σε θέματα τα οποία σχετίζονται με την εσωτερική αγορά Όπω επίσης και του κεκτημένου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε λοιπόν ένα σύστημα νομικό, το οποίο είναι πολύ στερεό για να εξασφαλίσουμε την ακαιρεότητα της εσωτερικής αγοράς. Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε πως δεν πρόκειται εδώ για διαπραγμάτευση ε, θεμάτων φορολογικών. Δεν καλύπτεται αυτό από την εντολή τη διαπραγματεύσεων. Οι χώρες αυτές ακολουθούν τους διεθνείς κανόνες του ΩΣΑ για την φορολογία. Αυτό έχει γίνει στο πλαίσιο των εργασιών μας ε, μαζί τους και έχουν βγει από τον κρίζο κατάλογο. Είναι πολύ θετικό αυτό. Οπότε, φιλοδοξία μας είναι να προχωρήσουμε ακόμα πιο πολύ με μια συμφωνία πλαίσιο για τις χώρες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μάρτενς, να σας πω πως η ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα γίνει 4 Φεβρουαρίου και Ολομέλεια 1η Μαρτίου. Τελευταία σημεία, στο πρώτο, στην πρώτη Ολομέλεια του Μαρτίου. Το επόμενο σημείο είναι η Συμφωνία Συνεργασίας και Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σιγκαπούρης στην ε, διάσκεψη 19 Οκτωβρίου του 2018 με την ΑΣΕΑΝ υπογράφηκε η συμφωνία αυτή και πέρασε από τις 8 Ιανουαρίου από το Συμβούλιο και ανακοινώθηκε ε, στο Κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα. Εμείς θεωρούμε ως Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων πως θα πρέπει να ε, τα δούμε όλα αυτά στα πλαίσια της συμφωνίας για την προστασία των εμπορικών μας συμφερόντων, όπως επίσης και συμφωνία για τις ελεύθερες συναλλαγές που έχουν υπογραφεί και αυτές τον Οκτώβριο με τη Σιγκαπούρη. Θέλουμε λοιπόν να σας παρουσιάσουμε αυτό το σχέδιο ψηφίσματος και συμφωνίες από τον κύριο Ιστούρης που ήδη το έστειλε στην Επιτροπή μας και μετά είχαμε 45 ε, τροπολογίες ε, οι οποίες μειώθηκαν και έχουμε 6 μεταβατικές τις οποίες αυτή τη στιγμή θα σας παρουσιάσει ο κύριος Ιτουρής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να σας πω πως έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Ευτυχώς τώρα η Σιγκαπούρη έχει συμμορφωθεί με όλα τα σημεία που είναι απαραίτητα για τις διαπραγματεύσεις και μετά από μια αυτή την μακρά περίοδο αναμονής έχουμε την έκθεση μπροστά μας. Λυπάμαι για τους σκιώδεις γιατί ήμουν λίγο σκληρός με το χρονοδιάγραμμα, με τις τροπολογίες και τα λοιπά, όμως ξέρετε είχαμε φιλόδοξο πρόγραμμα και δεν ξέρω αν ο συνάδελφος είναι εδώ για να τα πούμε. Α, να δούμε αν είναι εδώ η, η υπηρεσία εξωτερική δράση, είστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Να μειώσουμε λοιπόν τι προθεσμίε έτσι ώστε να εγκριθεί πριν το τέλο τη θητεία μα. Αυτό μα ζήτησε το Προεδρείο μα σήμερα, να κλείσουμε σύντομα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Οπότε είναι καλή συμφωνία, θα σα τα στείλω γραπτά και το μόνο που θέλω να πω είναι πω θα δημιουργηθεί μια μεικτή επιτροπή από εκπροσώπους σε υψηλό επίπεδο από όλα τα μέρη, έτσι ώστε να έχει η ε, σωστή εφαρμογή και καλή λειτουργία η συμφωνία αυτή. Και επίσης να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της ΑΦΕΤ και το Προεδρείο που με στήριξαν γιατί μείωσα τις προθεσμίες και τους συναδέλφους γιατί καταφέραμε ένα συνενετικό κείμενο που θα ψηφίσουμε αύριο, ε, το οποίο και στην ψηφοφορία αύριο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά, και για την ε, παρουσίαση, αλλά κυρίω για τη συντομία με την οποία την ολοκληρώσατε. Ο κύριος Μάρτιν έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και θα προσπαθήσω και εγώ να είμαι σύντομο. Ξεκινώ ευχαριστώντα τον εισηγητή για την πολύ καλή συνεργασία που δεν ήταν δεδομένη, όπως είπατε και εσεί. Ε, Όμω καταλήξαμε σε καλέ συμβαστικέ λύσει που θα καταθέσουμε αύριο για ψηφοφορία στην Επιτροπή. Αυτή η συνεργασία, λοιπόν, αυτή η συμφωνία συνδέσης και συνεργασία είναι θετική και για τις ε, σχέσεις μας με την κοινότητα ΑΖΕΑΝ εν γέννη, για να αναπτυχθούν οι σχέσεις μας μαζί τους. Αντίστοιχα με τις ε, συμφωνίες θερικής οικονομικής σχέσεις που έχουμε με την Ινδονησία, το Βιετνάμ κτλ. Αλλά και για να αναπτύξουμε διμερείς ε, σχέσεις με την κυβέρνηση της Συγκαπούρης ώστε να συζητήσουμε θέματα όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον, κλιματική αλλαγή, φορολογικά. Που θα αντιλαμβάνονται οι συνάδελφοι ότι αυτή η συμφωνία συμπληρώνει την, την συμφωνία περί επενδύσεων και τη συμφωνία περί ελεύθερων συναλλαγών. Άρα έχουμε πολύ καλύτερε σχέσει με την ε, Σιγκαπούρη. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ενισχύσουμε και τον διάλογο σε τρεις τομείς, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα των ΛΟΑΔΜΑ και θανατική ποινή με στόχο βέβαια την κατάργησή τη. Και θα συνεχίσουμε τις επαφές ε, με την Σιγκαπούρη ώστε να επιδιώξουμε βελτίωση των συνθήκων και λακωνικά, σε σχέση βέβαια και με τόσο είπαμε πριν με, τα μικρο, με τις μικροχώρες, ε, θα εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι σε μία επιστολή η Ιδονησία δεσμεύεται να συνεργαστεί στην αυτόματη ανταλλαγή δεδομένων φορολογικών και τραπεζιών. Τραπεζικών ευχαριστώ. Τάνοκ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον παλιό φίλο και συνάδελφο Αντώνιο Λόπες. Ήμουν παρόν σε διαπραγματεύσεις. Η ομάδα μου υποστηρίζει συμβαστικές τροποβουλίες Συμφωνώ με το όσο είπε ο David Μάρτιν για την ε, προστασία όχι μόνο της, Ευρω... της σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Σιγκαπούρη αλλά που κυμαίνεται γύρω από το εμπόριο και τα οικονομικά αλλά και αυξάνοντας το πεδίο ε, και την αντανάκλαση και στις σχέσεις με τις άλλες χώρες ΑΣΕΑΝ που πιστεύω μπορεί κάποια στιγμή να προχωρήσουν σε επίπεδο τελωνιακής ένωσης. Είναι χώρα βέβαια και της Βρετανικής Κοινοπολιτείας σε Σιγκαπούρη. Είναι τραγική ηρωνία το ότι ορισμένοι ή πολλοί από αυτούς που ψήφισαν για τον Brexit θεωρούν ότι με την απαχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα αναβιώσει η κοινοπολιτεία ενώ πολλέ χώρες κοινοπολιτείες και σημαντικές, όχι μόνο η Σικαπούρη, αλλά και η Αυστραλία, ο Καναδάς και άλλες ετοιμάζονται να υπογράψουν τα συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς την ώρα που το Ηνωμένο Βασίλειο ετοιμάζεται να αποχωρήσει από αυτήν. Είναι πολύ θλιβερό λοιπόν αυτό και επίσης με την ευκαιρία ήθελα να πω ότι πολλοί από τους πιο σκληροπυρηνικούς του Brexit θεωρούν ότι ε, η απορρίθμιση που επικρατεί οικονομικά σαν σύστημα στη Σιγκαπούρη θα ήταν το καταλληλότερο και για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την ε, αποχώρηση του από την Ηνωμένη Ευρώπη. Ωστόσο εδώ έχουμε να κάνουμε στη Σιγκαπούρη δηλαδή με ένα σύστημα κανόνων και περιορισμών που καθόλου δεν μοιάζουν με ένα σύστημα τύπου Far West, όπως ορισμένοι φαίνεται να θέλουν. Στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ αυστηρά ρυθμιζόμενη η οικονομία. Είναι ενδιαφέρον εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλούς λόγους η Σιγκαπούρη. Και πιστεύω ότι θα ενισχυθεί περισσότερο η θέση του με τις συμφωνίες αυτές. Θα υποστηρίξουμε λοιπόν την έκθεση στην ψηφοφορία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Τάνοκ και τελευταία θα δώσω το λόγο στην εκπρόσωπο της ΕΙΕΦ, την κυρία Άμπρα Λογκάτη, που είναι αρμόδια για τις διεθνείς σχέσεις και τις σχέσεις με το Βιετνάμ και τη Σιγκαπούρη. Σας ε, θέρμα παρακαλώ, όχι παραπάνω από 2-3 λεπτά. Α, καλώς, έχετε δικαίωμα και να με μιλήσετε. Απλώς σας είχα στον κατάλογο γι' αυτό. Εγώ υπέβαλα μία ερώτηση. Η ΑΕΔ συμφωνεί να επισπεύσουμε τη διαδικασία γιατί έλα, ε, λάβατε επιστολή από τον πρόεδρο της ε, ΑΦΕΤ. Υπάρχει βούληση και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επισπευστούν τα πράγματα για να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό αυτή η συμφωνία. Μήπως μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση του εισηγητού. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Η ΕΕΔ ήδη έχει ε, διαβιβάσει το Δεκέμβριο στο Συμβούλιο το σχετικό έγγραφο. Και από ό,τι ξέρω το Συμβούλιο στις 8 Ιανουαρίου το διαβίβασε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε και εμεί είμαστε ιδιαίτερω πρόθυμοι να προωθήσουμε τη διαδικασία σύντομα. Και φυσικά θεωρούμε ε, χρήσιμη την ενίσχυση των σχέσεων με τη Σιγκαπούρη. Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με του προλαλήσαντε. Ε, έμεινε ικανοποιημένο ο εισηγητής μα, Λαμπρά. Θα ψηφίσουμε αύριο στην Επιτροπή μας την έκθεση αυτή και στις 11 με 14 στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ και τους διερμηνείς, τους και τις διερμηνείς για την υπομονή τους και τους ευρωβουλευτές που τηρήσαν το χρόνο τους. Ραντεβού αύριο σε 9 με τις ψηφοφορίες.